Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Ας ξεκινήσουμε να ζητήσω τους φίλους που βρίσκονται εδώ από τον τύπο να καθίσουν. Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζάς, τον Μάριο Ντράγκη, για τον τρίτο νομισματικό διάλογο του 2015. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για μας ε, το να ακούσουμε τις, από το στόμα του τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας η οποία χαρακτηρίζεται από μια επιβράδυνση στις ε, ε, οικονομίες των αναδυόμενων οικονομιών όπως στην Κίνα ειδικότερα, οπότε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις προοπτικές ε, οικονομίες ε, από τον κύριο Ντράγκη, τις ευρωπαϊκές προοπτικές ε, και τι αναμένεται για την οικονομική ανάκαμψη που λέγεται ότι αναμένεται να συνεχίσει να επιταχύνεται αλλά λίγο πιο αργά. Θα μάθουμε επίσης ποια είναι η οικονομική στάση αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, το ζήτημα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το ευρύτερο ζήτημα βελτίωσης ε, της διακυβέρνησης της νομισματικής ένωσης στο πλαίσιο της έκθεσης των πέντε προέδρων. Πολλά λοιπόν σημαντικά ζητήματα. Τη Δευτέρα Είχαμε επίση μια ενδιαφέρουσα προπαρασκευαστική συνάντηση για τον νομισματικό διάλογο που συζητήθηκα μεταξύ άλλων η διάδραση μεταξύ νομισματικής ε, πολιτικής και ε, μακροπροληπτικής πολιτικής. Ε, οπότε αναμένω να μας πει κάτι και γι' αυτό ο κύριος Ντράγκη. Και φυσικά μετά θα ακολουθήσει ένας γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Κύριε Ντράγκη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε έκτακτες και εξαιρετικές προκλήσεις. Καταρχήν είχαμε την ε, μακροσκελή και περίπλοκη συζήτηση για το νέο πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας. Και τώρα σε ένα θέμα που βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουμε την πρόκληση να περιθάλψουμε ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων που χρειάστηκε να ξεριζωθούν από τις αιστείες τους. Και τα δύο αυτά γεγονότα, παρόλο που διαφέρουν πολύ στη φύση τους, έδειξαν και πάλι ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή μόνο εν τη ενώση με βάση την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Και αυτό είναι το δίδαγμα που θα, πρέπει να αντλήσουμε και για τις μελλοντικές μας προκλήσεις. Στις σημερινές μου παρατηρήσεις και σχόλια θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο βασικά θέματα. Καταρχήν, τις εκτιμήσεις μας για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις συνέπειες τους στα ζητήματα της νομισματικής πολιτικής και δεύτερον, τις προτάσεις που υποβάλαμε από κοινού με τους συναδέλφους στην έκθεση των πέντε προέδρων. Και ξεκινώ με το πρώτο θέμα. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση των οικονομικών εξελίξεων από την τελευταία κρόση που είχαμε τον Ιούνιο. Το καλοκαίρι η βιομηχανική παραγωγή και άλλοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας έδειξαν σημάδια προσαρμοστικότητας. Ταυτόχρονα, το μακροοικονομικό περιβάλλον έγινε όλο και πιο δύσκολο και απαιτητικό. Οι προβλέψεις μας, ε, οι μακροοικονομικές του Σεπτεμβρίου, έδειξαν μια στενέστερη οικονομική ανάπτυξη και χαμηλότερη αύξηση των ποσοστών πληθωρισμού από αυτά που αναμέναμε στις αρχές του έτους. Το ποσοστό του πληθωρισμού θα μείνει κοντά στο μηδέν στο εγγύς μέλλον, πριν αρχίσει να ξανανεβαίνει κατά τα τέλη του έτους. Θα χρειαστεί όμως περισσότερος καιρός από ό,τι φανταζόμασταν προηγουμένως για να επανέλθει και να σταθεροποιηθεί σε επίπεδα γύρω στο 2%. Η επιβράδυση της οικονομικής ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες, ένα ισχυρότερο ευρώ και η μείωση των πετρελαϊκών τιμών και των τιμών των βασικών προϊόντων είναι οι κυριότερες αιτίες των εξελίξεων αυτών. Ως εκ τούτου, ε, ναι, η κίνδυνοι μείωση ε, της ανάπτυξης ε, και του πληθωρισμού έχουν γίνει ορατοί. Για πολλές από τις αλλαγές αυτές είναι λίγο πρόωρο να κρίνουμε με σιγουριά αν θα αποκλίνουν από την αρχική πορεία που περιμέναμε να ακολουθήσει ο πληθωρισμός όταν αποφασίσαμε να διευρύνουμε το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων τον Ιανουάριο. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να προσδιορίσουμε κατά πόσο η μείωση της ανάπτυξης που διαπιστώσαμε στις αναδυόμενες οικονομίες είναι προσωρινή ή μόνιμη και να εκτιμήσουμε τις αιτίες της μείωσης της διεθνούς τιμής βασικών προϊόντων, καθώς και τα πρόσφατα επεισόδια σοβαρών χρηματοοικονομικών αναταράξεων. Ως εκ τούτου θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς ε, όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα λαμβάνουμε και τις συνέπειες που θα έχουν στις προβλέψεις για τη σταθερότητα των τιμών. Τα μέτρα νομισματικής μας πολιτικής μαζί με τα TLTRO, στι στοχευμένε μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης, εξακολουθούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο κόστος και τη διαθεσιμότητα των δανείων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Μέχρι στιγμή έχουν αποσοβήσει μια ε, με, καταμετρημένη ε, επιδείνωση των οικονομικών συνθήκων παρά τη, στην πραγματική οικονομία παρά την αύξηση της χρηματοοικονομικής αστάθειας και η σταθερή μείωση του κόστους δανεισμού ενισχύει την εγχώρια ζήτηση, στηρίζοντας ε, την κατανάλωση αναλώσιμων αγαθών και δίνοντας ε, κίνητρα για τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό καθιστά την ε, οικονομία της Ευρωζώνης πιο ανθεκτική στις εξωτερικούς κραδασμούς. Αν όμως πραγματοποιηθούν οι κίνδυνοι μείωσης του πληθωρισμού και μεσοπρόθεσμα και μάλιστα πιο δραστικά από ό,τι υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση. Το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων έχει αρκετή εγγενή ελαστικότητα και ευελιξία. Θα προσαρμόσουμε το μέγεθος, τη σύνθεσή του και τη διάρκεια του, όπως αν χρειαστεί, και αν ε, γίνει απαραίτητη περισσότερη όθηση από πλευράς νομισματικής πολιτικής. Γνωρίζω ότι παρακολουθείτε το, εκ του σύνεγγυς ε, το πιθανό αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οι συντονιστές της ΕΚΟΝ επέλεξαν το θέμα αυτό ως ένα από τα θέματα της σημερινής συζήτησης. Οπότε συνεχίζοντας ε, αυτά που είπα και το Μάρτιο, θα ήθελα να επισημάνω ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες του κινδύνους στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι υπαρκτή αυτή η κίνδυνη επί του παρόντος. Αν κάτι τέτοιο παραστεί αναγκαίο και καταστεί εμφανέ, η μακροπροληπτική πολιτική και όχι η νομισματική πολιτική θα είναι το εργαλείο που θα επιλέξουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτού του κινδύνους. Εδώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πρόσφατη εμπειρία μας ό,τι αφορά τα σχετικά εργαλεία. Τα τελευταία δύο χρόνια οι εθνικές αρχές στην Ευρώπη δραστηριοποιήθηκαν στη θέσπιση και εφαρμογή μακροπρο, μακροπροληπτικών πολιτικών, όπως ανώτατα όρια σε ε, δείκτες δανείου αξίας και χρέους εισοδήματος, προκειμένου να ενισχυθεί δομικά η αγορά ανυπόθηκων δανείων και ε, να μειώσουμε τις τιμές ε, ε, στα, στα στεγαστικά δάνεια. Επίσης, για να ισχυθεί το τραπεζικό σύστημα, οι χώρες έχουν εισάγει κάποιες προφυλακτήρες κατά των συστημικών κινδύνων, πέραν των ε, προστατευτικών μέτρων για τις ε, παγκοσμίως συστημικές τράπεζες και άλλες σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Αυτά λοιπόν τα μακροπροληπτικά εργαλεία έχουν καλύψει το δανεισμό μεταξύ των τραπεζών και είχαμε μία μετατόπιση ε, της χρηματοδότησης της οικονομίας προς τις ε, μη τράπεζες, μη τραπεζικούς θεσμούς. Γι' αυτό η κάλυψη του μακροπροληπτικού πλαισίου έχει, ε, αρχίζει να επεκτείνεται και στον, ε, στην παράλληλη ε, τραπεζική βιομηχανία, προκειμένου να, να, να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι του χρηματοοικονομικού κλάδου. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για την Ελλάδα. Στην ακρόση του Ιουνίου είχα ζητήσει μια περιεκτική και δίκαιη συμφωνία με την Ελλάδα. Τις επόμενες ε, εβδομάδες ε, μετά, ε, μετά τον Ιούνιο ακολούθησαν πολλές συζητήσεις και τεράστιες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκομένους. Αλλά είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί τελικά έγινε δυνατή η σύναψη της συμφωνίας. Και αν εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία αυτή, το νέο πρόγραμμα θα φέρει την Ελλάδα σε θέση ανάπτυξης και πάλι προκειμένου να αποκομίσει όλα τα ωφέλη της συμμετοχής στο κοινωνόμισμα. Η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με βάση τις διατάξεις του νομικού πλαισίου, συμμετείχε στη διαπραγμάτευση του προγράμματος. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολούθησε εκ του ε, την εφαρμογή τη διάταξη επίκουσα στήριξη ρευστότητα από την Τράπεζα τη Ελλάδα με βάση του κανόνε και λαμβάνοντα υπόψη την προοπτική μια ευόδοση ε, των διαπραγματεύσεων ε, σχετικά γρήγορα. Θα ήθελα τώρα να πω λίγα λόγια για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τι θα ακολουθήσει μετά την έκθεση των πέντε Προέδρων. Οι θερινές διαπραγματεύσεις ε, αποκάλυψαν και πάλι το γεγονός ότι το θεσμικό μας πλαίσιο δεν είναι αντάλογο ούτε αντάξιο των απαιτήσεων του κοινού νομίσματος. Στην έκθεση των πέντε προέδρων που δημοσιεύσαμε αμέσως μετά την τελευταία μας ακρόαση, οι πέντε πρόεδροι εστερνίζονται μία πεποίθηση. Το γεγονός ότι για να γίνει σταθερή και θαλερή η νομισματική ένωση, χρειαζόμαστε μια πληρέστερη ένωση. Και μάλιστα στην έκθεση δεν περιγράφουμε μόνο αυτή την κοινή μας πεποίθηση, αλλά υποβάλλουμε και ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη προκειμένου να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο στόχο. Ο οδικό αυτός χάρτη θα πρέπει να γίνει ο διζητή των επόμενων μηνών. Κατά τη δική μα γνώμη, δύο στοιχεία είναι ιδιαίτερη σημασία. Πρώτον, παρά όλες τις προσπάθειες των ενδιαφερομένων, η κρίση έδειξε ότι η Νομισματική Ένωση απαιτεί ένα πολιτικό κέντρο. Ένα κέντρο που θα μπορέσει να λάβει τις κατάλληλες δημοσιονομικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις για την Ευρωζώνη και μάλιστα με γρήγορο και διαφανή τρόπο, με πλήρη δημοκρατική νομοποίηση και μία δέσμη ευθυνών που θα λαμβάνει από τους νομοθέτες. Και υπό το πνεύμα αυτό έχω πευθύνει επανειλημμένως έκκληση για μια μετάβαση από τον συντονισμό που στηρίζεται στους κανόνες σε μια διανομή της κυριαρχίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η έκθεση μάλιστα προτείνει ένα, οικονομικό, ένα Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τέτοιου είδους ιδέες θα πρέπει να αναπτυχθούν αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και στις άλλες πολιτικές μας. Η έκθεση των πέντε προέδρων προσδιορίζει ότι η ΟΝΕ θα πρέπει να ενισχύσει και την εργαλειοθήκη της προκειμένου να διαχειριστεί και να αποτρέψει την ε, αύξηση χρηματοοικονομικών, ε, δημοσιονομικών και μακροοικονομικών κινδύνων. Τα τελευταία χρόνια με τις ε, μεταρρυθμίσεις ενίσχυση του πλαισίου ε, οικονομική διακυβέρνηση, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, λάβαμε σημαντικά βήματα προκειμένου να ενισχύσουμε την εργαλειοθήκη μα για την αποτροπή και τη διαχείριση των κρίσεων. Αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη πλήρω. Θα πρέπει ως ονούπο να ολοκληρώσουμε και την Τραπεζική Ένωση με ένα κοινό μηχανισμό στήριξης ε, για το ενιαίο Ταμείο Εξηγίας Τραπεζών και το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Και τα δύο αυτά στοιχεία χρειάζονται για να δημιουργήσουμε ένα γνήσιο ενιαίο τραπεζικό σύστημα αντάξιο του ενιαίου νομίσματός μας. Και φυσικά έτσι θα ενισχύσουμε την αξιοπίστεια της Τραπεζικής Ένωσης και θα υλοποιήσουμε την αρχική της υπόσχεση δηλαδή να ε, δια, διαρρήξουμε τον ε, δεσμό μεταξύ των τραπεζών και του δημόσιου χρέους, να καταστήσουμε το οικονομικό σύστημα πιο ευπροσάρμοστο και ανθεκτικό και να προσπίσουμε τα συμφέροντα των φορολογουμένων. Ταυτόχρονα, ξεπερνώντα τα όρια τη ε, τραπεζικής ένωσης και του τραπεζικού κλάδου, θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και στην ανάπτυξη της ένωσης των Κεφαλαίων Προκειμένου να διευρύνουμε το, το διασυνοριακό ε, ιδιωτικό θέμα της ανάληψης ε, κινδύνων. Επιπλέον θα πρέπει να αποφύγουμε τις ανισορροπίες, όποια μορφή και αν έχουν, ε, και να αποφύγουμε τη μετατροπή τους και την διεύρυνσή τους σε ένα περιβάλλον κρίσης. Χρειαζόμαστε μια νέα διαδικασία σύγκλησης που θα στηρίζεται στην ικανότητα της οικονομίας μας να αντέξει σε κραδασμούς και να τους ξεπεράσει το συντομότερο δυνατό. Αυτό προϋποθέτει όχι μόνο ένα στιβαρότερο χρηματοοικονομικό σύστημα, όπως είπα προηγουμένως, αλλά και ισχυρότερη διακυβέρνηση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αυστηρότερο έλεγχο των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. Για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν στους κραδασμούς, θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα στρώμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά μαζί θα αποτελέσουν τα βήματα ολοκλήρωσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να έχουμε μια ευρωζώνη, μια ευρωζώνη που θα επιβιώσει, αλλά που ταυτόχρονα θα είναι θαλερή και θα ανθίσει περαιτέρω. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Ντράγκη. Εκτιμώ ιδιαίτερα τα όσα είπατε για την ανάγκη καλύψης ε, με το ε, μακροπροληπτικό πλαίσιο το τομέα το τραπεζικό και συμμεριζόμαστε τις φιλοδοξίες σας ε, σε αυτό το θέμα. Περνάμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Να ενημερώσω τα μέλη ότι μετά από την απόφαση των συντενιστών θα εφαρμόσουμε τις νέες διευθετήσεις πολύ αυστηρά, οπότε δύο λεπτά αυστηρά για τις ερωτήσεις και μετά αν μείνει χρόνος μετά από τις απαντήσεις θα ε, αφήσουμε και επιπλέον πέντε λεπτά για τη συνέχιση. Πρώτος ομιλητής. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, δείξατε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, ε, με τα οποία μπορούμε βέβαια να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτησή μας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δείξω εγώ ένα θέμα το οποίο αφορά εμάς, τη δική μας την πολιτική ομάδα, κυρίως το ΕΛΚ, κάτι που απασχολεί το ΕΛΚ. Συγκεκριμένα λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέβαλε και αυτή τα μάλα έτσι ώστε να περιορίσει τις αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και εδώ αναφέρομαι κυρίως σε χώρες με υψηλό χρέος και μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Μέχρι τώρα λοιπόν μιλάμε για χώρες οι οποίες από πλευράς οικονομικής δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι η μεγαλύτερες. Όμως ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου, επιπτώσεις έστω και από αυτές τις χώρες είναι απρόβλεπτες. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, κατά την άποψή μου, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί εάν χαλαρώσουμε τα δημοσιονομικά κριτήρια. Εσείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχετε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο σας δεσμεύει, άρα δηλαδή καταλήγουμε στο ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει πρέπει να αποκτήσουν σταθερότητα, ότι πρέπει να μειωθεί το χρέος των κρατών αυτών και να επιβληθούν, να εισαχθούν αν θέλετε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ξεκινώντας λοιπόν η συζήτηση θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς ως ΕΚΤ πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε εκείνους οι οποίοι επιδεικνύουν κάποια ολιγορία κατά την εφαρμογή του, ε, συμφων... του Συμφώνου Σταθερότητας. Και μόνο αυτό, αλλά μερικοί μιλούν και για χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, ακριβώς το επισημένο αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, μόλις ε, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του ε, οδικού χάρτη, του χάρτη πορείας, όσον αφορά την περαιτέρω ολοκλήρωση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, καταφύγαμε σε όρους από την, ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλώντας για μια πιο τέλεια ένωση, a more perfect union. Για να συνεχίσουμε λοιπόν το ταξίδι μας χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Και για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη πρέπει να σεβόμαστε και τους κανόνες που βάζουμε μόνοι μας στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα επέλθει περαιτέρω ολοκλήρωση που ε, θα επιδεικνύει μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε κοινού θεσμού αν δεν επαναφέρουμε την αξιοπιστία. Η σταθερότητα και το σύμφωνο ανάπτυξης είναι μόνο ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζονται ξανά από σταθερότητα. Υπάρχει ένα γενικότερο θέμα που αφορά στη βελτίωση της ικανότητας να μπορεί κανείς να στέκεται μόνος του στα ίδια του τα πόδια. Πριν λοιπόν συμφωνήσουμε και καταλήξουμε σε κοινό δρόμο, κοινή πορεία για να επιμερίζουμε κινδύνους οι οποίοι θα μπορούσαν να πλήξουν διάφορους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προϋπάρξει αυτό που σας είπα. Έχετε αν θέλετε χρόνο για να επανέλθετε με την ερώτησή σας. Όχι, η κυρία Φερέρα. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε για τόσα είπατε επίσης. Είπατε σημαντικά πράγματα τα οποία απασχολούν και εμάς πρωτίστως. Η πρώτη μου ερώτηση σχετίζεται με τον πρώτο τομέα που αναφέρατε. Έχετε κάνει ό,τι μπορούσατε για να σώσετε το ευρώ και το έχετε σώσει μέχρι στιγμής. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εξωτερικό περιβάλλον το οποίο επιβραδύνεται σιγά σιγά το πρόβλημα της Λατινικής Αμερικής, της Κίνας, ε, η Fed ε, που δεν ε, αύξησε τα επιτόκια. Οπότε για πόσο χρόνο μπορούμε να σταθούμε στην Ευρώπη με μόνο τις δικές μας πολιτικές κατά της κρίσης χωρίς να περάσουμε σε κάποιο είδους δημοσιονομική πολιτική όπως εσείς έχετε ζητήσει επανειλημμένως η πρόταση σας ε, στην έκθεση των πέντε πρόεδρων να υπάρχει κάποιο κοινό ε, στοιχείο, ένα κοινό Υπουργείο Οικονομικών, αυτό θα πάρει χρόνο. Οπότε ποιο είναι το όραμά σας για το εγγύς μέλλον. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω αφορά την ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε τη διαδικασία και στη μέση του δρόμου να πούμε δεν θέλουμε να το πάμε παραπέρα. Είναι ένα παιχνίδι. Επιχνίδι επικίνδυνο, αλλά το οποίο θα σώσει την Ευρώπη. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που αποτελούν τροχοπέδι και ε, στα οποία μπορεί να βοηθήσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο να αρθούν ε, εγγύσεις ας πούμε για τις καταθέσεις, για τις ε, ελάχιστες καταθέσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες ανεξαρτήτως χώρας όπου βρίσκονται. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που θα βοηθήσει την εμπιστοσύνη. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν για ποιο λόγο διστάζουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει και αρχίζουμε να αμφισβητούμε και να αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι σωστό αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως είπα προηγουμένως, η μείωση της ανάπτυξης έχει αυξήσει φυσικά τον κίνδυνο ε, μείωση τη ε, ύφεση ε, παρότι είναι πρόμοιο να πούμε κάτι τέτοιο. Αυτή η μείωση είναι μόνιμη ή απλά προσωρινή, δεν γνωρίζουμε. Πολλές όμως προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αναδυόμενες οικονομίες αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να εξαφανιστούν άμεσα. Δεδομένου αυτού του περιβάλλοντος, η απλα προσωρινη δεν γνωριζουμε πολλε ομως προκλησεις που εχουν να αντιμετωπισουν οι αναδυομενε οικονομιες αυτη συνεχίζεται στην Ευρωζώνη. Παρότι λίγο πιο αργά. Όχι πολύ πιο αργά παρεπιπτόντως, διότι έχουμε αναθεωρήσει τις προβλέψεις μας και αναμένουμε ότι για το υπόλοιπο του έτους, βάσει των στοιχείων που έχουμε σήμερα, τα οποία το επιβεβαιώνουν αυτό, αναμένουμε ότι το υπόλοιπο του έτους θα συνεχίζει με έναν τέτοιο χαμηλότερο δίκτυο ανάπτυξη ε, του δεύτερου τριμήνου αλλά είμαστε σε επαγρύπνηση για πιθανούς κινδύνους και η νομισματική μας πολιτική θα ασκηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε εφόσον χρειαστεί. Η ανάκαμψη λοιπόν συνεχίζει να υποστηρίζεται από τις χαμηλές πετρελαϊκές τιμές από την χωρία νομισματική μας πολιτική που προσαρμόζεται στις συνθήκες. Αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι για να μετατραπεί η ανάκαμψη από κυκλική σε διαρθρωτική. Οι χώρες πρέπει να προβούν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή εμείς λέμε ότι η νομισματική πολιτική βοηθά και βοήθησε πράγματι και θα έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε για ποιο λόγο βοηθά, πώς γίνεται και βοηθά την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μόνη της. Δεν μπορεί να μετατρέψει μια κυκλική ανάκαμψη σε διαρθρωτική. Για να γίνει αυτό, οι χώρες πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Στοιχείο κλειδί αυτή τη εξυγίανση και τη παγίωση τη ανάκαμψη είναι η επαναφορά τη εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη έχει πολλά πρόσωπα, πολλά πτυχές. Υπάρχει εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές που τώρα έχει επανέλθει μετά το 2012 κατά βάση. Παρατηρείται συνεχής βελτίωση όσον αφορά την εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αλλά όπως είπα προηγουμένως η εμπιστοσύνη βασίζεται και σε άλλα στοιχεία. Ένα από τα οποία είναι η γενικότερη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι οι τρέχοντες κανόνες τηρούνται, αλλά και εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι το μοντέλο, το πρότυπο, η ατζέντα περαιτέρω ολοκλήρωσης ε, ε, έχει ληφθεί στα σοβαρά πραγματικά και ότι γίνονται συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπιστοσύνη επίσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι δεσμεύσει θα εφαρμοστούν όπως η δέσμευση ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης που είναι παρούσα και τώρα πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να αναμένουμε ε, ουσιώδεις ε, συνθήκες, ε, αλλαγές στις συνθήκες πριν ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Αυτή η υπεποίθηση χρειάζεται για να επανέλθει η εμπιστοσύνη και αυτή ζητείται όταν αναφερόμαστε σε τήρηση των κοινών κανόνων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μεριάς. I will Greek. Αρκετοί ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συχνά αναλαμβάνει δράσεις οι οποίες εξέρχονται των ορίων της εντολής της όπως αυτή προσδιορίζεται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι καταρχάς τις επιστολές που έστειλε ο κύριος Τρισέ προς τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας υπό το πρόσχημα της δίθεν διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Στην περίπτωση της Ελλάδας οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ στην άσκηση οικονομικής πολιτικής γίνονται μέσα από τη συμμετοχή της ΕΚΤ στην Τρόικα. Όμως η συμμετοχή της ΕΚΤ στην Τρόικα οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων, καθώ έτσι αναιρείται η ανεξαρτησία τη ΕΚΤ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η Τρόικα δρά υπό την πολιτική καθοδήγηση του Eurogroup. Ήδη από τι αρχέ του 2015, ο Γενικό Εισαγγελέα του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γνωμοδότησή του στην υπόθεση OMT, επισήμανε ότι προκειμένου να θεωρηθεί ένα μέτρο εντασσόμενο στην νομισματική πολιτική τη ΕΚΤ, ένα πρόγραμμα όπω το OMT, η ΕΚΤ τότε οφείλει να απέχει από κάθε είδου παρέμβαση στα προγράμματα χρηματοδοτική βοήθεια που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ESM ή του EFSF όπω ακριβώ συμβαίνει με την Ελλάδα. Δηλαδή, ο Γενικό Εισαγγελέα σα ζήτησε με άλλα λόγια να φύγετε την Τρόικα. Στη συνέχεια το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Ιουνίου στην απόφασή του δέχτηκε τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα και επισήμανε ότι όταν η ΕΚΤ προβαίνει στην αγορά κρατικών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές πρέπει να συνοδεύει τις παρεμβάσεις της με αρκετές εγγύσεις. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2015 δέχτηκε τροπολογία που υπέβαλα με την οποία ζητούσα την έξωση της ΕΚΤ από την Τρόικα σας ερωτώ λοιπόν κύριε ντράγκη πότε σκοπεύει η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να φύγει από την τρόικα προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής ένωσης να πάψει να βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων και να σταματήσει να εφαρμόζει το σκληρό μνημόνιο 3 που φτωχοποιεί παραπάνω τον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε, ε, λυπάμαι πάρα πολύ. Η ΕΚΤ δεν έχει πει τίποτα από όλα αυτά. Και δεύτερον, η ΕΚΤ ε, δεν πρόκειται να παραμείνει στην Τρόικα για πάντα. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Τώρα είμαστε σε περίοδο κρίσης, αλλά η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή απλά εφαρμόζει τους νόμους. Δεν είναι θέμα της ΕΚΤ αν θα φύγει από την Τρόικα ή όχι. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επισημάνω στον κύριο Ντράγκη ότι ίσως θα πρέπει να διαβάσει ξανά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαβάσει ειδικότερα την παράγραφο 102 η οποία λέει επιλέξει εντεύθεν έπεται ότι όπως και ο Γενικός Εισαγγελέας επισήμανε στο σημείο 227 των προτάσεων του ότι όταν η ΕΚΤ προβαίνει στην αγορά κρατικών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές πρέπει να συνοδεύει τις παρεμβάσεις της με επαρκείς εγγύησεις. Και οι εγγύησεις αυτές περιγράφονται από τον ίδιο το Γενικό Εισαγγελέα στο σημείο 227 και σε άλλα σημεία των προτάσεών του που σας λέει ότι δεν μπορείτε να είστε ταυτόχρονα μέλος της Τρόικας και να ασκείτε νομισματική πολιτική με προγράμματα τύπου OMT επομένως θα πρέπει να δείτε το θέμα αυτό κύριε πρόεδρε Thank διότι εσείς τη συμμετοχή της Thank you. Otherwise there is no time for the answer. This, the, the follow-up cannot be unlimited. I will, I will take... No, no, please, Mr. President Draghi. It was very clear the point. Ήταν σαφές το θέμα. Δεν έμεινε πολύ σκέλο για την απάντηση. Η τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα OMT. Μπορεί αργότερα να τα πούμε κατηδίαν, αν θέλετε, για να δούμε αν συμφωνούν οι αναγνώσει που κάνουμε τη απόφαση. Η κυρία Σιλβί Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε και ευχαριστώ για το έργο σας στην έκθεση των πέντε Προέδρων. Νομίζω ότι στείλατε ένα μήνυμα εμπιστοσύνη σε μια κρίσιμη στιγμή και ένα μήνυμα εμπιστοσύνη προ το μέλλον. Αναφερθήκατε και στο ζήτημα της εξωτερικής εκπροσώπησης, της εξωτερικής ε, εκπροσώπησης ε, της Ευρωζώνης, ε, το άρθρο 138 της Συνθήκης. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Γιούνκερ. μάλιστα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω έκθεση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Έχω μια ερώτηση λοιπόν σχετικά. Χρησιμοποιώντας τη λογική που διέπει την έκθεση των πέντε προέδρων, τι μπορούμε να κάνουμε Βραχυπρόθεσμα πρόθεσμα και ποιοι είναι οι κοινοί μας μακροπρόθεσμοι στόχοι. Αν προσπαθήσουμε βραχυπρόθεσμα πρόθεσμα να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να μας, κάνει, να μας πει περισσότερα τι κάνει στην Επιτροπή της ε, Βασιλείας ή στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Γιατί η Τραπεζική Ένωση αφορά τις ε, ε, σχέσεις μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε σε θέματα συνεργασίας μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Επίσης, μέσω πρόθεσμα, πολύ σωστά μιλήσατε για εκδημοκρατισμό των οργάνων της Ευρωζώνης. Ε, εκδημοκρατισμό σημαίνει κοινοβουλευτικός έλεγχος, ενώ μιλούμε για εξωτερική εκπροσώπηση από το Eurogroup. Ενώ ο πρόεδρος του δεν θεωρεί ότι είναι υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς βλέπετε λοιπόν τη λογοδοσία της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωζώνης είναι ε, θέμα κρατικό και ε, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει, όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχουμε εμεί ανεξάρτητη γνώμη. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική, είναι σαφές ότι η εξωτερική εκπροσώπηση ανήκει στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Συμβούλιο ε, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή στην Επιτροπή της, Βα... της Βασιλείας, ξέρετε ότι συμμετέχουμε και στα δύο όργανα, και ως ΕΚΤ και στα πλαίσια του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού και εκεί μεταφέρουμε τις απόψεις μας στους διεθνείς οργανισμούς. Αλλά και πάλι και τα κράτη-μέλη είναι μέλη και των οργανισμών αυτών. Και αυτή τη στιγμή, αλλά και στο παρελθόν, αυτό που προσπαθούμε είναι να διαμορφώσουμε κοινέ απόψεις εντός της Ευρωζώνης για τα θέματα που συζητώνται. Μερικές φορές τα καταφέρουμε να έχουμε τέτοια κοινή γνώμη ενία και άλλες φορές όχι. Αυτό δεν μας εμπόδιζε όμως να καταλήξουμε σε συμφωνία για πολλά θέματα, συμφωνία που τελικά ικανοποίησε όλα τα κράτη-μέλη. Πάντως, αν ρωτάτε μια τεχνική κρίση ή αξιολόγησή μου κατά πόσο επιδέχονται βελτιώσει αυτά τα πράγματα, η απάντηση είναι καταφατική. Τώρα, τι είδου βελτίωση εννοούμε, αυτό θα εξαρτηθεί από εσά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Εσεί θα αποφασίσετε. Δευτερολογία. Παρά είστε μετριόφρον. Γιατί συμμετέχετε στην έκθεση των πέντε προέδρων. Δίνετε τη γνώμη σας για ιδιαίτερα πολιτικά ζητήματα. Θα ήθελαν όχι σήμερα να δούμε κάποια στιγμή πώς θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για το τι συμβαίνει στην Επιτροπή της Βασιλείας ή στο FSB, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ευχαριστώ. Αν ε, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή ΕΚΟΝ για τη θέση της ε, στους οργανισμούς αυτούς ε, αλλά και στους υπόλοιπους οργανισμούς νομίζω ότι από αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Είμαστε έτοιμοι. Ο κύριος Φάβιο κύριε Ντράγκη, αν κατάλαβα καλά, η ΕΚΤ έχει αναθέσει εξωτερικές νομικές μελέτες ε, σε σχέση με την ε, αιτιολόγηση της ε, μη αποδοχής περαιτέρω ελληνικών ομολόγων ως εγγυήσεων στις αρχές του χρόνου. Θα μπορούσατε να κοινοποιήσετε αυτές τις μελέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Δεύτερον, αναφέρεται ότι ο κίνδυνος μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης όπως αρκετά έχει αυλυνθεί. Ε, τι ρόλο πιστεύετε ότι θα παίξει μια μεταρρύθμιση των τραπεζών για τις μακροπροληπτικές ε, πολιτικές στην Ευρώπη, για παράδειγμα διαχωρισμός ορισμένων επενδυτικών ε, τραπεζικών δραστηριοτήτων από τις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες λιανικής και επίσης ήθελα να ρωτήσω κάποια ειδήσει που ακούμε στα μέσα δείχνουν ότι ορισμένοι Ορισμένα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ υποφέρουν από burnout. Ε, με ποιο τρόπο φροντίζει η ΕΚΤ ε, διασφαλίζει ότι τηρούνται οι όροι της σχετικής οδηγίας, ε, υπολογίζεται τις υπερορίες και πώς. Και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η εκτεχή εισάγει διαιτές ανώτατο όριο για κάποιες ε, θέσεις ε, προσωπικών ε, στην ΕΚΤ και για ποιο λόγο δεν διασφαλίζει την ίση αμοιβή μετά από εννέα μήνες. Για να απαντήσω στην τρίτη ερώτηση, επανεξετάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα, κάνουμε τη δική μας έρευνα, έρευνα προσωπικού, την έρευνα της ΕΚΤ, ε, προχωρούν ταυτόχρονα και όλα αυτά τα ζητήματα προσωπικού βρίσκονται υπό συζήτηση αυτή τη στιγμή με το προσωπικό μας. Για τη δεύτερη σας ερώτηση δεν είμαι ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο. Κοιτάω τα πράγματα ως έχουν και ε, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών είναι ένα παράδειγμα όπου πρέπει να προχωρήσουμε ώστε οι δομές μας να γίνουν πιο ανθεκτικές, ισχυρότερες και ικανές να αντέχουν κραδασμούς. Οι τραπεζικές αυτές λοιπόν μεταρρυθμίσεις, οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και το ζήτημα εκεί είναι ότι δεδομένου το τραπεζικό μας σύστημα διαφέρει σημαντικά από εκείνο άλλων χωρών, το βασικό ζήτημα είναι πώς θα προβούμε σε μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος όπου θα προχωρήσουμε προς τη δημιουργία ισχυρότερων ε, ε, ιδρυμάτων ε, διαχωρίζοντας ενδεχομένως τις δραστηριότητες λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του δικού μας τραπεζικού συστήματος και διασφαλίζοντας ότι οι, τράπεζε, οι τραπεζές μας δεν θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές όπου πραγματοποιούνται διαφορετικού τύπου τραπεζικές μεταρρυθμίσεις. Οπότε η μεταρρύθμιση αφήνει κάποιο περιθώριο ε, διακριτικής ευχέρειας στους εθνικούς ε, ε, επόπτες για να περάσουν τις θέσεις τους. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτή η μελέτη μη αποδοχή των ελληνικών ομολόγων, αλλά εδώ μου δίνεται ευκαιρία αναθεώρησης της τρέχουσας κατάστασης. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος ε, στην Ελλάδα, τόσο δημοσιονομικά όσο και όσον αφορά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Τώρα ε, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το τρίτο πρόγραμμα και συνεχίζουμε, ε, συνεχίζονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το ζήτημα είναι θα επαναφέρουμε την αποποίηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα την εξαίρεση. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εντάσσεται η χώρα σε ένα πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής βοήθειας. Πρέπει να συμμορφώνεται με αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι και αυτό που συνέβη στην πορεία των τελευταίων μερικών εβδομάδων και θα συνεχίσει να συμβαίνει με τις επόμενες εβδομάδες. Πρέπει ουσιαστικά να είναι ιδιοκτήτης του προγράμματος ε, μέσω όλων πολλών διαφορετικών κυβερνήσεων και πρέπει να συμμορφώνεται με τις ε, δράσεις προτεραιότητας, δηλαδή αποδεικνύοντας ότι είναι διοκτήτης του προγράμματος μέσω ε, αποφασισμένων δράσεων που σε αυτό το πρόγραμμα αφορούν δημοσιονομική πολιτική, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και άλλες σημαντικές ε, αποφάσεις πολιτικής. Αφού αυτό επιτευχθεί, απομένει ένα βήμα. ουσιαστικά η αξιολόγηση αυτής της βιωσιμότητας. Όπως γνωρίζετε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέφρασε ανησυχίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Αλλά αν γίνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ε, βάσει ενός σημαντικού προγράμματος που θα παράγουν ανάπτυξη αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη, δημοσιονομική βιωσιμότητα και οικονομική ε, βιωσιμότητα και υπάρξει ιδιοκτησία αυτού του προγράμματος, τότε το περιθώριο χαλάρωσης ε, ανακουφίσης του χρέους ε, θα γίνει υπαρκτό, το οποίο είναι σημαντικό ε, για να κριθεί και η βιωσιμότητα του χρέους. Όταν όλα αυτά αποτελούν γεγονός, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έχει τους δικούς του κανόνες. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάποια ζητήματα, κάποια όρια εκδοτό, εκδοσής και φυσικά δεν μπορούμε να αγοράζουμε ομόλογα ενώ πραγματοποιείται αναθεώρηση. Οπότε όλα αυτά ε, μας λένε ότι ας προχωρήσουμε ε, γρήγορα, ας υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, ας ε, εφαρμόσουμε τις δράσεις προτεραιότητας και ας ολοκληρώσουμε επιτυχώς την αναθεώρηση. And I don't know whether this was a confidential information, but I still would like to see them. Εγώ είμαι ρωθικά για τις μελέτες. Δεν ξέρω αν είναι πιστευτικές προφορίες, αλλά θέλω να τις δω. Ernest Urtasun. Ernest Urtasun. Thank you, Chair, Mr. Draghi. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, θα ήθελα να επιμείνω λιγάκι στην Ελλάδα και στις αποφάσεις που Στην πρώτη απόφαση που ελήφθη μετά τον Ιούλιο είπατε ότι παρότι οι ελληνικές τράπεζες είναι τυπικά βιώσιμες και φερέγγιες, η ΕΚΤ εφαρμόζει μια δυναμική αξιολόγηση η οποία αμφισβητεί την φερεγγιότητα αυτών των τραπεζών και ε, δημιουργείται το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Αυτό οδήγησε στο ότι το Συμβούλιο δεν αύξησε τον ΕΛΑ και τις αποφάσεις για τον ΕΛΑ. Όμως σε τουλάχιστον μία περίπτωση στην Κύπρο και πριν από τον bailout ο ΕΛΑ αποδείχθηκε ως ένας μηχανισμός ο οποίος έσωσε μία τράπεζα, τότε όμως υπήρχαν στοιχεία ότι η τράπεζα ήταν αφερέγγια. Και παρότι κρίθηκε ότι ήταν αφαιρέγγια, η τράπεζα διασώθηκε. Η ερώτησή μου λοιπόν κύριε Ντράγκη είναι η εξής. Από τέτοια διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάμεσα στους ε, θεσμούς ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αμφισβητείται το θέμα της ε, αφαιρεγγιότητας, ότι η αξιολόγηση αφαιρεγγιότητας δεν είναι απαραίτητη προπόθεση για να αυξηθεί ο ΕΛΑ, αλλά το Συμβούλιο μπορεί αυθαίρετα να ορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ΕΛΑ αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και θα ήθελα επίση κύριε Ντράγκη να γνωρίζω κατά πόσο πιστεύετε ότι οι κανόνε για τον Έλα είναι σαφεί ή όχι, λαμβάνοντα υπόψη αυτά που είπα. Και το τελευταίο που θέλω να πω κύριε Ντράγκη είναι το εξή. Ε, είχατε ασκήθηκε έντονη κριτική στις αποφάσεις για την Ελλάδα γιατί ε, ήταν πολύ στενά συνδυασμένες με την ε, Ευρωζώνη. Πιστεύετε παρόλα αυτά ότι η τράπεζα πραγματικά αμφισβητήθηκε κυρίως κατά το μήνα Ιούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απαντήσω σύντομα στο πρώτο ερώτημα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ασυμμετρία. Δηλαδή, βασιστήκαμε στην αξιολόγηση της ε, εποπτικής αρχής περιαφερεγγιότητα. Στην Κύπρο ήταν κεντρική τράπεζα και στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν ο νέος μηχανισμός σταθερότητας, ο SSM. Όσον αφορά τον έκτακτο μηχανισμό των ΕΛΑ, εκεί είμαστε σαφείς. Οι κανόνες του ΕΛΑ ποτέ δεν προβλέπουν ότι η χορήγηση ρευστότητα ε, είναι χωρίς προϋποθέσεις και η χορήγηση γίνεται χωρίς κανένα όριο όπως ε, μας ασκήθηκε η κριτική. Ούτε ποτέ έχει λεχθεί ότι το θέμα της ρευστότητα των τραπεζών είναι δυναμικό όπως είπαν και κάποιοι άλλοι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι και αυτοί άσκησαν κριτική. Φτάνω λοιπόν στην απάντησή μου για το τρίτο ερώτημα. Κοιτάξτε, το να έχει κάνει κριτική και από δεξιά και από αριστερά, αυτό τι σημαίνει ότι η ΕΚΤ επικρίνεται διότι δεν έκοψε τον ΕΛΑ πολύ πολύ νωρίς και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε τον ΕΛΑ να τον κατεβάσει στο μηδέν, να... Ε, το χέψι, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και κάποια άλλη στιγμή που διατηρήθηκε όλα, δεν μειώθηκε, αλλά διατηρήθηκε σε αυτό το επίπεδο και πάλι δέχτηκε κριτική. Άρα δηλαδή, όποια και αν είναι κριτική, εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος σε σχέση με αυτά που πράττει η ΕΚΤ. Αν έχω χρόνο, θα ήθελα να κάνω μία ε, δεύτερη απάντηση. Όχι, δεν έχετε δυστυχώ, διότι το σύνολο είναι 5 λεπτά, δύο για την ερώτηση και τρία για την απάντηση. Περνάμε στον επόμενο ερωτώντα, τον κύριο David Κόμπορν Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να υποβάλω διαδικαστικό πριν να περάσω στο δίλεπτο που δικαιούμαι για την ομιλία μου. Τι διαδικαστικό, γρήγορα. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 55 εκατομμύρια ευρώ ε, κοινό κεφάλαιο στο, στην ΕΚΤ, αλλά δυστυχώς κλείνει το μικρόφωνο του κύριε Κόμπερ. Μα δεν είναι διαδικαστικό αυτό κύριε Κόμπερ. Περάστε στην ερώτηση κατευθείαν. Ξεκινάει το δίλεπτό σα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει, θέ, δεν έχει έδρα, ε, δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη, στην ΕΚΤ. Δεν θα πρέπει να υφιστάμεθα δηλαδή τις συνέπειες ε, της ύπαρξής της. Ο κύριος Φλάναγκαν από την Ιρλανδία δεν είναι στην Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να ρωτήσει τον κύριο Δράγκη, τον πρόεδρο της ΕΚΤ, γιατί δεν ήρθε στην Ιρλανδική Βουλή για να συζητήσει του σοβαρούς ισχυρισμού ότι η ΕΚΤ ήθελε, απείλησε να χρεοκοπήσει την Ιρλανδική οικονομία για να μην και ήθελε ουσιαστικά ε, να μετακυλήσει τις ζημίες των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών στις Ιρλανδικές και στους Ιρλανδικούς φορολογουμένους. Και μην ξεχνάμε τι έγινε ε, μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τι χρειάστηκε να αναλάβουν οι Γερμανοί φορολογούμενοι. Ε, ο κύριος Φλάνεγκα δεν είναι μέλος της Επιτροπής ΕΚΟΝ, αλλά ακριβώς επειδή επλήγει από τη δράση της ΕΚΤ ο Ιρλανδικός Λόγος, πιστεύω ότι πρέπει να του δώσουμε το λόγο για να σχολιάσει αυτό που θέλει να ρωτήσει. Μπορείτε να του δώσετε χρόνο από την ομάδα σας, αν θέλετε. Ναι, αλλά δεν είναι μέλος της ομάδας μας. μη με διακόπτετε, κύριε Κόμπερν. Για το Ιρλανδικό θέμα έχουμε την απόφαση των συντονιστών να συμπεριλάβουμε αυτό το ζήτημα στην επόμενη ε, συνάντηση που θα έχουμε τον, ε, του νομισματικού διαλόγου. Τον Νοέμβριο εκεί θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε το ζήτημα. Αυτή είναι η απόφαση των συντονιστών. Το ελλανδικό ζήτημα θα μπει στο νομισματικό διάλογο του Νοεμβρίου. Μη με διακόπτετε κύριε Κόμπερν. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Κόμπερν. Μην διακόπτετε τη συνεδρίαση παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Κόμπερν. Ρωτήστε τον κύριο Ντράγκη. Μα οι συντονιστέ συμφώνησαν ε, και μάλιστα είπε ο κύριο Δράκη στην Ιρλανδική Βουλή ότι είναι υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφωνήσαμε το θέμα αυτό το Ιρλανδικό να το συζητήσουμε στο νομισματικό διάλογο του Νοεμβρίου. Επόμενο ομιλητή τώρα ο κύριο Μπερνάρ Μονό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δραγκή παρατηρώ στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάποια αντίφαση. Θέλουμε κάποιες εξηγήσει. Αφενός ε, υποστηρίζεται την οικονομική ανάπτυξη, τον έλεγχο των επιτοκίων που βρίσκονται στο χαμηλότερο ιστορικό επίπεδό τους και με τη χρήση μη συμβατικών ε, εργαλείων των LTROs, του ELA και την ποσοτική χαλάρωση του 2015 με σκοπό να δοθούν κίνητρα στις τράπεζες να δανείζουν στην πραγματική οικονομία και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από πληθωρισμό που μας εξηγήσετε πέρσι. Πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να πείτε ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν πάνε καλά παρότι ο στόχος της πολιτικής σας ε, είναι καλός. Επίσης ε, Θέλετε μεταρρύθμιση της προληπτικής ε, κατάστασης των ε, κρατικών ομολόγων. Ε, αυτό βελτιώνει τη φερεγγιότητα των τραπεζών και τη ρευστότητά τους, αλλά επιδεινώνει την κατάσταση των κρατών. Υπάρχει κίνδυνος σχετικός με αυτά που μπορεί να επιδεινωθεί. Έτσι λοιπόν με τον καιρό η ρευστότητα θα υπονομευτεί και θα υπονομεύσει και τη δυνατότητα των τραπεζών να πάρουν και άλλους κινδύνους, δηλαδή δανεισμού. Και έτσι οι αγορές ε, θα μπορούν να επηρεάσουν έμεσα την οικονομική πολιτική των ε, εκδοτριών χωρών ασκώντας πίεση στις τράπεζες. Πώς εξηγείται την αντίφαση αυτή μεταξύ των στόχων. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίφαση σε αυτό που λέτε. Ε, είναι ευέλικτη η νομισματική μας πολιτική και θα συνεχίσει να είναι η ίδια βάσει της εντολής μας η οποία λέει ότι το ποσοστό πληθωρισμού θα πρέπει να είναι κοντά αλλά κάτω από το 2% και εμείς ε, είμαστε μακριά από αυτόν τον στόχο αυτή τη στιγμή. Οι πολιτικές μας λειτουργούν, ξέρετε, διότι παρότι οι προοπτικές ε, της παγκόσμιας οικονομίας φαίνονται ζωφερές ε, βάσει της ε, αρχής της ομιλίας μου υπάρχουν και κάποιες θετικέ εξελίξεις από πιστοτική πλευρά και θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε αυτές στις θετικέ εξελίξεις στην Ευρωζώνη. παρατηρείται ανάκαμψη των πιστοτικών αγορών, η οποία συνεχίζεται ακόμη και σήμερα και γίνεται όλο και πιο έντονη. Όλες οι έρευνες που έχουμε διεξάγει και στις τράπεζες και δηλαδή στην πλευρά των δανειστών και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πλευρά δηλαδή των δανειολήπτων ε, όπως φαίνεται ε, έχει αυξηθεί η ποσότητα των δανείων όχι μόνο ποσοτικά αλλά και όσον αφορά την έκτασή τους δηλαδή η δανειοδότηση έχει αυξηθεί και στις χώρες που αντιμετωπίζουν πιο δύσκολες συνθήκες και στις υπόλοιπες. Τα ποσοστά δανεισμού έχουν μειωθεί. Χρησιμοποιούμε αυτό που ονομάζεται ε, σύνθετος ε, δείκτης κόστους δανεισμού το οποίο δείχνει ότι τα ποσοστά δανεισμού, τα επιτόκια δανεισμού έχουν μειωθεί κατά 7 ε, πόντους από βάσεις ε, από τότε που ανακοινώθηκαν ε, τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και βλέπουμε ότι και το χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρών δανειοληπτών έχει μειωθεί τόσο σε θέματα ποσότητας όσο και σε θέματα κόστους. Συνολικά λοιπόν αυτές οι εξελίξεις στις πιστοτικές αγορές φαίνεται να ενισχύουν την εντύπωση ότι συνεχίζεται η ανάκαμψη Μιλάμε για σταδιακή ανάκαμψη, όχι για κάτι απότομο και ξαφνικό και μεγάλου μεγέθους. Ωστόσο, συνεχίζει και προχωρά προς το καλύτερο. Αυτό με την πολύ αργή ε, βελτίωση των αγορών. Αυτές είναι οι θετικές πτυχές της ανάκαμψης και αυτό είναι η διαφορά με το παρελθόν ότι όλα αυτά καθοδηγούνται κυρίως από την εγχώρια κατανάλωση. Οπότε κατά μία έννοια αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές μας φέρνουν αποτέλεσμα. Κατά πόσο υπάρχει αντίφαση με τις εποπτικές μας πολιτικές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλετε να θέσετε ουσιαστικά. Να σας εξηγήσω λίγο με γενικούς όρους και με τα πιο συγκεκριμένα για το θέμα που αναφέρατε εσείς για τα κρατικά χρέη και τα κρατικά ομόλογα και την αξιολόγηση επικινδυνότητάς τους σε γενικές γραμμές, υπό γενικούς όρους, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ μιας προσαρμοστικής νομισματικής πολιτικής και της στενής επιτήρησης του τραπεζικού συστήματος. Εάν μια τράπεζα ε, βρίσκεται σε αδύναμη θέση και δεν διαθέτει κεφάλαιο, δεν πρόκειται να δανείσει. Εάν μια τράπεζα ε, έχει επενδύσει τα περιουσιακά της στοιχεία σε επικίνδυνα ε, προγράμματα δεν θα δανείσει. Συνεπώς απαιτείται ισχυρή εποπτική δράση ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ανάκαμψη θα συνοδεύεται από ένα ισχυρό πιστοτικό σύστημα. Αυτά λέει και η εμπειρία μας από το 2010-2011 και σχεδόν ολόκληρο το 2012 όταν τα πάντα από μακροοικονομικής πλευράς και από πλευράς νομισματικής ε, πολιτικής ε, υπήρχαν για να δώσουν όθηση στην ανάπτυξη με σοβαρή επέκταση της ρευστότητα και παρόλα αυτά το τραπεζικό σύστημα δεν παρήχε πιστώσεις στην οικονομία. Έχουμε περάσει αυτό το σκόπλο γιατί, διότι οι τράπεζες ε, ενδυναμώθηκαν πολύ σημαντικά πριν και μετά από την ε, ολοκληρωμένη αξιολόγηση του SSM. Και τώρα βλέπουμε ότι οι πιστώσεις σημειώνουν αυξητική τάση και όταν αναφέρομαι σε ισχυρή εποπτεία πρέπει να βασίζεται αυτή σε γεγονότα ρεαλιστικά σε μια ψύχρεμη αξιολόγηση του κινδύνου οπότε η ισχυρή εποπτική δράση δεν έρχεται σε αντίφαση με την προσαρμοστική νομισματική πολιτική ουσιαστικά αποτελεί προϋπόθεση για αυτή, ώστε αυτή η νομισματική πολιτική να μπορέσει να έχει πραγματικά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία. Ε, θα το συζητήσουμε... Ε, εγώ είχα πει να το συζητήσουμε ούτως ή άλλως. Θα ήθελα εγώ να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά την απογοήτευση που νιώθω βλέποντας τις αντιδράσεις κάποιων κρατών μελών που δεν είναι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένα και που ενδεχομένως ε, θα συνεχίσουμε να έχουμε μία κλιματική προσέγγιση όσον αφορά την ε, ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Λοιπόν, η ερώτησή μου προς εσάς αφορά το European Deposit Insurance Scheme, το θέμα το, της εγγύησης των καταθέσεων. οι τράπεζες θα έχουν ε, κάποια backstop, κάποια εγγύηση, απόθεμα δικό τους, αλλά εσείς θεωρείτε ότι αν τελικά συστηθεί αυτό το ταμείο και ε, συνδυαστεί με το Ταμείο Διάσωσης τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω έχει σχέση με την νομισματική πολιτική. Νομίζω ότι μια χαλαρή νομισματική πολιτική κάποια μέρα ε, θα πρέπει να ε, προσαρμοστεί ανάλογα με την ανάπτυξη. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι το να έχουμε μια σφιχτή νομισματική πολιτική αυτό απαιτεί μια πρωτοφανή προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ ποιοι είναι οι κίνδυνοι της ε, νομισματικής σας πολιτικής ε, την εποχή που έχουμε χαμηλά επιτόκια. Το θέμα της δημοσιονομικής προσαρμογής ε, και των τραπεζών. Πώς ακριβώς τα κρίνεται όλα αυτά, απάντηση του κυρίου Ντράγκη. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, απαιτεί να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση του προγράμματος εγγύησης των καταθέσεων και θα πρέπει να ε, συσταθεί και να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο Διάσωσης, Single Resolution Fund. Τα κράτη-μέλη όταν συνέστησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβαν αυτές τις αποφάσεις. Κατά τα άλλα, δεν είναι σωστό κατά κάποιον τρόπο να με ρωτάτε περισσότερο για τις οικονομικές και λιγότερο για τις πολιτικές επιπτώσεις. Ε, υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχουν όμως και υποχρεώσεις οι οποίες έχουν αναλυφθεί και οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Το πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εγγύησης Καταθέσεων βεβαίως και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα έναντι των εθνικών αντίστοιχων προγραμμάτων. Πρώτον, θα ενισχύσει τα προγράμματα αυτά και δεύτερον, οι στόχοι της ε, πολιτικής μας των μεταρρυθμίσεων τα πέντε χρόνια ήταν να χαλαρώσουν τα σχέδια ανάμεσα στις τράπεζες και τους οφειλέτες. Τώρα λοιπόν έχουμε μία εποπτική αρχή, έχουμε ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης και έτσι λοιπόν τις τράπεζες παντού τις αντιμετωπίζουμε στο ίδιο επίπεδο. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για τους καταθέτες. Γιατί να μην αντιμετωπίζεται και αυτή με τον ίδιο τρόπο ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τίθεται θέμα αρχής. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εσείς με ρωτήσατε για την ε, έξοδο από αυτή τη νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται τώρα. Κοιτάξτε, έχουμε τα εργαλεία και εγώ θα ήθελα απλά να πω ότι το πρόβλημα πράγματι υφίσταται. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε κύριε Ντράγκη που ήρθατε. Βέβαια, είναι όντως πρωτοκλασσά το πρόβλημα και είναι πρόωρο να μιλούμε τώρα για έξοδα από τέτοια νομισματική πολιτική. Έχω δύο ερωτήσεις. Ο οικόνομης αυτής της εβδομάδας είχε τη φωτογραφία του Τζέρεμι Κόρμπιν που επαναφέρει το εργατικό κόμμα στη δεκαετία του 60. Δεν είναι και πολύ δίκαιο αυτό, είναι μάλλον άδικο. Γιατί ποιο πολιτικό ηγέτης μιλούσε για τέτοια θέματα στη δεκαετία του 60, την ποσοτική χαλάρωση. Αλλά ο, ο κύριος Κόρμπιν ζήτησε ποσοτική χαλάρωση για τον κόσμο, όχι για τις τράπεζες. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη. Γιατί συμφωνούν μαζί του ακόμη και κάποιοι οικονομολόγοι. Αυτό είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Αν και, και στο Κοινοβούλιο ε, ακούστηκαν αυτέ, αυτές οι ιδέες. Γιατί να μην χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάποιε επενδύσει από το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Επίση, ο William Μπάουτερ είπε, αν η Citibank ε, έχει προβλέψεις για ύφεση και αν θέλουμε ε, μάνα εξ ουρανού, όχι ποσοτική χαλάρωση ε, για τους ανθρώπους, τότε να δούμε τι θα γίνει με την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Χαίρομαι που είπατε ότι είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα και της ποσοτικής χαλάρωσης και της αγοράς περιουσιακών στοιχείων. το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου το πρόγραμμά σας συμβάλλει και, συμβάλλει και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η απάντηση στη τελευταία ερώτηση είναι καταφατική. Το πρόγραμμά μας είναι όντως αποτελεσματικό και θα φανούν τα πλεονεκτήματα με το χρόνο. Καταρχήν ο δανεισμός ανακάμπτει και ακόμη και στις ε, χώρες που έχουν ε, βρεθεί σε δύσκολη θέση ε, αρχίζει και διαφαίνεται κάποια οικονομική ανάπτυξη μετά από αρκετά χρόνια. Γίνεται νέος δανεισμός υπάρχει ανάκαμψη της πίστης και μιλούμε για καθαρές ροές εδώ. Δηλαδή, μικτές ροές μείων ε, ε, εξυπηρέτηση προηγούμενων δανείων. Είναι βέβαια σταδιακή, επαναλαμβάνω, αυτή η πρόοδος. Αργή, αλλά σταθερή. Και υπάρχει αυτή η πρόοδος ε, σταδιακή, γιατί σε μερικές περιπτώσεις έχουμε κόκκινα δάνεια που επιβαρύνουν το ισοζύγιο των τραπεζών. Και επιδεινώνουν τον νέο δανεισμό. Αλλά υπάρχει μια αργέλα σταθερή πρόοδος. Και μάλιστα φάνηκε μέχρι στιγμής η αποτελεσματικότητα του προγραμματός μας. 387 ε, δισεκατομμύρια έχει φτάσει το TLTRO, στοχευμένες μακροπρόθεσμες πράξεις αναχρηματοδότησης. Και έχουμε αποδείξεις ότι αυτοί που ε, είχαν περισσότερη πρόσβαση στο πρόγραμμα είναι αυτοί που δάνεισαν περισσότερο και μάλιστα δάνεισαν περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εκεί τα επιτόκια δανεισμού ήταν που μειώθηκαν περισσότερο. Οπότε έχουμε ενδιαφέροντες συσχετισμούς μεταξύ των προγραμμάτων μας και των αποτελεσμάτων, της αποτελεσματικότητάς τους. Δεύτερη παρατήρηση. Για εκατοντάδες χρόνια οι κεντρικές τράπεζες ε, μεταβίβαζαν κονδύλια κεφάλαια στην οικονομία είτε μέσω των τραπεζών είτε μέσω των αγορών. Αυτά γνωρίζουμε για τις ενέσεις κεφαλαίου από τις κεντρικές τράπεζες. Οπότε τέτοιες ιδέες ε, συζητώνταν ανέκαθεν και παντού. Και εμείς συμμετέχουμε στις συζητήσεις αυτές και σε πανεπιστημιακούς κύκλους και σε άλλα φόρα. Επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και κάποιες νομικές πτυχές που ισχύουν ε, για την Ευρωζώνη και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν αυτό το μάνα εξ ουρανού, αυτά τα, τα χρήματα που ρίχνουν από το ελικόπτερο συνάδουν με τη συνθήκη. Δεν θα πρέπει όμως έτσι να προεξοφλούμε οποιαδήποτε απόφαση. Πάντως η σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα απαιτεί να χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς και τις γνώσεις μας. Και αυτή τη στιγμή οι γνώσεις μας αυτές είναι. Ο κύριος Σάλμπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ κύριε Πρόεδρε μαζί σας ότι η εμπιστοσύνη έχει πρωταρχική σημασία για να παγιώσουμε και να εδραιώσουμε την οικονομική ανάκαμψη. Και επίσης σας συμφωνώ ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να μετατρέψει την συγκυριακή ανάκαμψη σε μια διαρθρωτική ανάκαμψη που θα είναι και βιώσιμη αλλά με απασχολεί η αστάθεια και η αβεβαιότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις αγορές. Καταρχήν, η αβεβαιότητα λόγω τη αμερικανική νομισματική πολιτική. Μερικοί εμπειρογνώμονε λένε ότι αυτή επηρεάζει περισσότερο τι τρίτε χώρε. Πολύ περισσότερο από ότι αύξηση των επιτοκίων. Επίση, υπάρχει η αβεβαιότητα λόγω τη αστάθεια της κινέζικης αγοράς. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Πιστεύετε ότι η αβεβαιότητα θα διαρκέσει για πολύ καιρό ακόμη. Και δεύτερον, αν συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα, φαντάζομαι ότι εσείς ε, θα συνεχίσετε την ποσοτική χαλάρωση, το QE. Αν συνεχιστεί όμως η αβεβαιότητα, αποκλείεται να χρειαστεί να λάβετε και κάποια πιο φιλόδοξα μέτρα νομισματικής πολιτικής ή κάποια πιο επιθετικά μέτρα νομισματικής πολιτικής. Γιατί πρόσφατα ακούσαμε ποιες θα ήταν ποια θα ήταν τέτοια μέτρα. Αποκλείεται δηλαδή να λάβετε και επιπρόσθετα πιο φιλόδοξα, πιο επιθετικά μέτρα νομισματικής πολιτικής σε περίπτωση που παραταθεί αυτή η αβεβαιότητα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι εδώ και καιρό βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι νομισματικές πολιτικές βρίσκονται σε αποκλίνοντα μονοπάτια ακολουθούν αποκλίνουσες κατευθύνσεις ανά τον κόσμο. Σε άλλες χώρες η ανάκαμψη προχωρεί και ενισχύεται και σε εμά, για παράδειγμα, η ανάκαμψη συνεχίζεται, αλλά είναι σταδιακή, είναι αργή, είναι σε πρόωρα, πρώιμα στάδια. Και μιλούμε για προβλέψεις μεσοπρόθεσμες σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό που έχουν προσαρμοστεί προς τα κάτω για τις μακροοικονομικές προβλέψεις. Οπότε αυτή η αβεβαιότητα είναι υπαρκτή. Η δεύτερη σας ερώτηση. Ρωτήσατε σε ποιο βαθμό αυτή η αβεβαιότητα θα προτρέψει την ΕΚΤ να αναλάβει κάποια μέτρα νομισματικής πολιτικής. Αυτό που έχω πει επανειλημμένος είναι ότι αν η αβεβαιότητα είναι λόγος της αστάθειας, και αν αυτή η αστάθεια δημιουργήσει επιδείνωση των χρηματοοικονομικών ε, συνθήκων και επιδεινωθούν και οι προβλέψεις μας, οι μεσοπρόθεσμες, τότε θα τη δράσουμε, θα αναλάβουμε δράσεις. Και όπως σας είπα, πολλές δράσεις τέτοιες είναι πιθανές. What can... May I? Yes, a very brief question. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Τι είδου δράσεις, αν αποφασίσετε να αντιδράσετε, θεωρείτε ότι πρέπει να λάβετε. Ε, ξέρετε, η σημερινή μας νομισματική πολιτική, η κοινή μας νομισματική πολιτική, θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματική. Οπότε παραμένουμε σε αυτήν πριν αρχίζουμε να εξετάζουμε τον δεχόμενο άλλων δράσεων αλλά όπως είπα είμαστε έτοιμοι και υπάρχει βούληση και ικανότητα να δράσουμε εφόσον χρειαστεί. Και όπως είπαμε το πρόγραμμά μας, ε, οι προβλέψεις μας ε, βασίζονται στην πλήρη υλοποίηση αυτού του προγράμματος που θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο και αν χρειαστεί θα ε, το προχωρήσουμε και πέρα του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ, Πέτρη Ζήμων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολλές συζητήσεις ε, με μικρές ε, περιφερειακές τράπεζες καταδεικνύουν ότι κατά τη δική τους άποψη η πολιτική επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τους δημιουργεί προβλήματα. Υπάρχουν οι δαπάνες, διακόπτεται ομιλητής, υπάρχουν και έμεσες δαπάνες, οι άμεσες και έμεσες δαπάνες, οι οποίες επιβαρύνουν τις ε, μικρές τράπεζες πολύ περισσότερο από τις μεγάλες τράπεζες. Οι μεγάλες τράπεζες έχουν 10-15 συνεργάτες ε, για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα, αυτές τις δαπάνες το κόστος διεκπαιρέωσης. Εσείς λοιπόν πώς μπορείτε να εμποδίσετε το ότι έχουμε αυτή την πολιτική επιτοκίων που δημιουργεί προβλήματα στις μικρές τράπεζες, από την άλλη όμως έχουμε ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος που δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα προκύψει μία κρίση η οποία οφείλεται ακριβώς σε αυτό το αίτιο το οποίο προκαλεί η ίδια Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω όσον αφορά τη ρύθμιση, ε, τη ρύθμιση regulation ε, ε, που εμείς συμβάλαμε πάρα πολύ αλλά και εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατότητες για μικρές και μεσαίες τράπεζες παραδείγματο χάρη στην περίπτωση ε, μικροδανειδητήσεων όπου πάνω από 25.000 ε, δάνεια για να δοθούν αυτά πρέπει να συμπληρωθούν ε, πάρα πολλά τετραγωνίδια. Εδώ είχαμε το συνάδελφό σας και εσάς πάρα πολλές φορές και μας είπατε ότι στο θέμα αυτό θα υπάρξουν διευκολύνσεις για τις μικρομεσές επιχειρήσεις. Όμως δεν διευκρινίστηκαν αυτές οι διευκολύνσεις και θέλω να ρωτήσω εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις από αυτού. Θα ήθελα να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Η τρέχουσα νομισματική πολιτική είναι αυτή που είναι, διότι έχουμε την εντολή της ε, νομισματικής σταθερότητας μέσω μακροπρόθεσμα κάτω από 2%. Αυτή είναι η εντολή μας. Η εντολή που μας έχει δοθεί δεν είναι να διασφαλίζουμε ότι οι τράπεζες θα είναι κερδοφόρες. Έτσι λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δηλαδή δεν θα αυξήσουμε τα επιτόκια γιατί κάποιες μικρές τράπεζες σε κάποια μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόβλημα με τα κέρδη τους. Βεβαίως ε, και έχουμε πρόβλημα ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται κάποιο θέμα ε, δημοσιονομικής αστάθειας αλλά αυτό πάλι μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εργαλεία. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι σχετικά με το project Anna Credit διότι έχει σαν στόχο να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα δάνεια και η χορήγηση δανείων. Τώρα, το ότι υπάρχουν κάποια τμηματικά στοιχεία που αφορούν αυτό το πρόγραμμα και το ότι είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Άρα δηλαδή εδώ μιλάμε για βασικές κεντρικές λειτουργίες που υπάρχουν σε όλους σε τις σωστά εύρυθμα λειτουργούσες τάξης πραγμάτων. Το πρόγραμμα αυτό το Credit, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη χορήγηση δανείων σε διάφορους οφειλέτες, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα ξέρουμε τι συμβαίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις τράπεζες γιατί έχουμε έρευνες και η Επιτροπή έχει τις δικές της τις έρευνες. Όμως θα ήταν ε, πραγματικά κάτι διαφορετικό το να έχει κανείς πραγματικά δεδομένα και νομίζω ότι θα βοηθούσε αυτό ε, σε σχέση με τις δανειοδοτήσεις, άρα δηλαδή θα οδηγούσε σε διεύρυνση των εγγύησεων, των collaterals που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την νομισματική πολιτική. Θα βοηθούσε στο να βαθμολογεί και να διαβαθμίζει κανείς καλύτερα το θέμα των εγγύησεων, δηλαδή θα βοηθούσε να τιμολογούμε, να αξιολογούμε τους κινδύνους, το ενδεχόμενο της, των haircuts, αλλά αυτά με βάση στοιχεία. Όλα αυτά θα έδιναν επίσης τη δυνατότητα να υπάρξουν και οικονομικές έρευνες. Ξέρετε, οι γνώσεις που έχουμε στην Ευρωζώνη είναι πολλές, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Οφείλουμε να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα για τις οικονομίες μας την περίπλοκη δομή τους, την πολυμορφία τους. Εμείς ε, δουλεύουμε συνεχώς για να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας. Και όταν θα το πετύχουμε θα ελέγχουμε καλύτερα τους κινδύνους δημοσιονομικής σταθερότητας. Όλα λοιπόν αυτά τα ωφέλη που θα συνεπάγεται αυτό το project βεβαίως και συνεπάγονται κόστος. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό το κόστος μπορεί να ε, ε, εκτιμηθεί με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα είναι αφόρητο το κόστος για τις περισσότερες τράπεζες. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Και κατά τα άλλα, ο ίδιος ο τραπεζικός τομέας θα επωφελείται επίσης από αυτό το project. Θα ήταν ε, λοιπόν ε, δυνατό να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες. Ε, οι τράπεζες θα μπορούσαν να έχουν περισσότερες δυνατότητες benchmarking γιατί θα μπορούσαν να λαμβάνουν υπόψη τους και την πραγματικότητα τραπεζικών φορέων και άλλων φορέων σε άλλες χώρες δεν χρειάζεται να σας πω ότι βεβαίως και πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό το project, ακόμα και αν είναι μεγάλο το κόστος. Αλλά σας είπα και πάλι θα προσαρμόσουμε το κόστος στις δυνατότητες ε, των τραπεζών. Ευχαριστώ Λούντα Μάγερ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που βρίσκεστε εδώ και εύχομαι ό,τι καλύτερο στο δύσκολο εγχείρημα που έχετε. Δύο ερωτήσει έχω. Κατά την ελληνική κρίση, πρώτον, η ΕΚΤ έπαιξε σημαντικό ρόλο σε κάποιε στιγμέ, διότι ουσιαστικά παρήχε τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Εκείνη την εποχή η, κυριαρχία των, η, συγγνώμη, η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών βασιζόταν στην προπόθεση ότι ε, θα γινόταν διαπραγματεύσει νέου προγράμματο από την ελληνική κυβέρνηση. Και η ερώτησή μου είναι Θεωρώ ότι αυτή ήταν μια πολύ πολιτική θέση της ΕΚΤ. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι σημερινοί κανόνες του ΙΕΛΕ είναι σωστοί. θα σας ε, ενοχλήσει αν ξαναμπείστε παρόμοια κατάσταση ΕΚΤ στο μέλλον. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την Κίνα. Η Κίνα ήταν μια οικονομία υψηλών επιδόσεων για ε, αρκετές ε, δεκαετίες και τώρα αποτελεί το αδύναμο σημείο της ε, παγκόσμιας οικονομίας εξάγοντα την επιβράδυνση και σε άλλες χώρες. Να σας ρωτήσω πρώτα πώς βλέπετε τις, την νομισματική πολιτική και την πολιτική, συναλλαγματική πολιτική ιδίω στην Κίνα και τις προσπάθειες τόνωσης της ανάπτυξης από την κινέζικη κυβέρνηση και δεύτερον σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι αυτό συμμορφώνεται με τη φιλοδοξία ε, της, ε, των κινέζικων αρχών να δουν το τους ως παγκόσμιο νόμισμα. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Σημειώνουμε. Ε, στη δεύτερη, συγγνώμη. Ε, θεωρούμε ότι η Κίνα, όπως και οι υπόλοιπες οικονομίες των G20, έχει δεσμευτεί στη, με τις συμφωνίες ε, G20 ε, όσον αφορά την ε, συναλλαγματική πολιτική. Και τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζονται στην Κίνα, όπως και σε άλλες περιοχές, οφείλονται και προσανατολίζονται προς στόχους της εγχώριας οικονομίας. Το γεγονός ότι επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τη συναλλαγματική ισοτιμία είναι απλά ένα αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, αλλά όχι πρωταρχικό του σκοπό. Δεδομένων αυτών, είναι σημαντικό η Κίνα να συνεχίσει την πορεία της και τι δράσει τη προς ε, ε, καλύτερη συναλλαξιμότητα και ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες που να καθορίζονται περισσότερο από την αγορά. Και είναι σημαντικό επίση η Κίνα να προβεί και να συνεχίσει τι ε, διαφορετικέ τη μεταρρυθμίσει. Για την πρώτη ερώτηση, αρνούμε ότι οι αποφάσει για το ELA είναι πολιτικής φύσης. Να επαναλάβω, επιτρέψτε μου, το λόγο. Το ELA είναι βοήθεια ρευστότητα που δίνεται σε φερέγγια ιδρύματα που έχουν επαρκείς ε, εγγύησεις. Οι εγγύησεις των ελληνικών τραπεζών είναι ως επιτοπλίστων ελληνικά, ελληνική τίτλη, ελληνικά ομόλογα. Οι αποφάσεις λοιπόν οικονομικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης επηρεάζουν την αξία αυτών των ομολόγων, δηλαδή τις εγγύσεις, δηλαδή και την απόφασή μας κατά συνέπεια να συνεχίσουμε ή να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το ELA. Αυτό που συνέβη είναι ότι για κάποιο χρονικό διάστημα οι, πολιτικές αυτές, οι αποφάσεις αυτές οικονομικής πολιτικής ήταν ε, εγκυτική αξία που βελτιωνόταν και μετά εγκυτική αξία που κατέστρεφε. Και έτσι αποφασίσαμε σε κάποια χρονική στιγμή ότι τα γεγονότα ήταν τέτοια που η αξία των εγγύσεων δεν ήταν επαρκής ώστε να αυξηθεί το ELA. Να σας υπενθυμίσω ότι αποφασίσαμε να μην μειώσουμε το ELA αλλά να το διατηρήσουμε σταθερό το οποίο παρεμπιπτόντως είναι το υψηλότερο που επιτέχθη ποτέ για οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωζώνη. Και μετά, όταν ελήφθησαν ε, αποφάσεις τέτοιες που ήταν δυνατή η ε, άρση αυτών των εμποδίων και οι αποφάσεις αυτές επηρέασαν, ε, επηρέασαν θετικά την αξία αυτής της εγγύησης, το ELA αυξήθηκε και δεν υπήρξε ένσταση ε, του Διοικητικού Συμβουλίου προς το αίτημα της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό δείχνει ότι η απόφαση δεν ήταν πολιτική. Ήταν απόφαση που βασίζεται στους κανόνες μας και οι κανόνες μας ουδέποτε έλεγαν ότι το ELA έπρεπε να είναι απεριόριστο και ανεφόρον. Επίσης, ουδέποτε είπαν οι κανόνες μας ότι οι αποφάσεις μας για την ρευστότητα των τραπεζών πρέπει να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται άμεσα και ότι εμείς μπορούμε να προβλέπουμε την μελλοντική του ε, ρευστότητα και φερεγγιότητα. Με λίγα λόγια, η ΕΚΤ δεν είναι ε, ο θεσμός που αποφασίζει το ποιο μέλο θα μείνει στην Ευρωζώνη και ποιο όχι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δρά και αποφασίζει θεωρώντας δεδομένο ότι όλα τα μέσα της ε, Ευρωζώνης θα συνεχίσουν να είναι μέλη της Ευρωζώνης. Άλλα θεσμικά όργανα έχουν την ευθύνη αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Περβάνος Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, εισαγωγική σας ε, ομιλία μιλήσατε για τη συζήτηση και την πρόταση για τη σύσταση ενός ε, Υπουργείου Οικονομικών της Ευρωζώνης. Ε, φαντάζομαι ότι κάτι προϋποθέτει και έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Μιλήσατε και για τη δημοκρατική ευθύνη. Ε, αυτά είναι αλληλένδετα κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να μιλούμε για κοινοβούλιο της Ευρωζώνης αν δεν συνδέεται άμεσα με έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Γιατί Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη δημοκρατίας. Είναι, επαναλαμβάνω, αλληλένδετες οι δύο έννοιες, αλλά και οι δύο χρήζουν αναθεώρηση των συνθήκων. Και όταν βλέπουμε τα όρια των δράσεών σας στα πλαίσια της νομισματικής πολιτικής που κάνατε βέβαια πάρα πολλά, αλλά έχουν και όρια οι δυνατότητές σας. Και κάποια στιγμή ανέκυψε και το θέμα της ε, δημοσιονομικής ικανότητας ε, και κάποιες ε, αντικυκλικές κινήσεις δεδομένη τη έκθεση ε, των πέντε Προέδρων, τη κατάσταση τη Ευρωζώνη, των προοπτικών, γιατί έχουμε το παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, αλλά έχουμε και την οικονομία των χωρών τη Ευρωζώνη. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, την πολυτέλεια του χρόνου μάλλον. Μήπως ε, πρέπει να σπεύσουμε με ταχύτερους ρυθμούς. Γιατί πολύ αργά πάμε. Στην αρχή έχουμε την ευθύνη, το αντικίνητρο και μετά το καρότο το κίνητρο. Ε, αλλά με, ίσως με τέτοια αργοπορία τελικά οδηγήσουμε στην καταβαράθρωση της Ευρωζώνης. Η, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο ξαναρχίζει τη συζήτηση για το χρέος και ιδιαίτερα το δημόσιο χρέος. Βέβαια, κάποιοι συνάδελφοι λένε πριν να ασχοληθούν με το δημόσιο χρέο, πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του πρώτα τα κράτη-μέλη. Μήπω όμω πιστεύετε ότι όταν έχουμε χαμηλό προϊθορισμό και χαμηλή ανάπτυξη, υπάρχει εγγενώ και ένα πρόβλημα κανόνων των κανόνων που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και κυρίως τις ε, υποχρεώσεις τους για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους τους. Συμφωνώ απόλυτα με το πρώτο σας σχόλιο. Κατά κάποιο τρόπο η έκθεση των πέντε προέδρων έχει το εξής μήνυμα. Υπάρχουν κάποιες βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν, αλλά δεν είναι μόνο οι βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις, γιατί αυτές οι βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις ανοίγουν το δρόμο και προλύνουν το έδαφος για μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και όραμα. Και το μακροπρόθεσμο όραμα έχει ε, αναπτύσσεται περισσότερο στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης, στους μακροπρόθεσμους στόχους και δεσμεύσεις. Δεν είναι καθόλου απλό το θέμα. Και εκεί θα ανακύψουν προκλήσεις. Το θέμα είναι, είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη πρώτα να υλοποιήσουν τις βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις τους και κατόπιν να παρουσιάσουν στους πολίτες τους και στους ψηφοφόρους τους ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα που θα συμφωνήσουν από τώρα και φυσικά θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να υλοποιηθούν όλα αυτά που προτείνονται στην έκθεση των πέντε πρόεδρων. Αλλά η πολιτική πρόκληση θα πρέπει τώρα να αναλυθεί, να αντιμετωπιστεί. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα και η βασική πρόκληση η οποία παρουσιάζεται στα κράτη-μέλη από την έκθεση των πέντε πρόεδρων. έχουμε χαμηλό πληθωρισμό, αλλά έχουμε και χαμηλά επιτόκια. Και αυτό για το δημόσιο χρέος έχει ε, εξισορροπητικό ρόλο. Και σε πολλές ε, χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, τα επιτόκια είναι κάπως μεταβλητά για το δημόσιο χρέος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες για το ποσοστό του πληθωρισμού, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να εξυπηρετούσουν το χρέος ε, το χρέος τους για τις χώρες που έχουν βιώσιμο χρέος είναι να αναπτυχθούν με ποσοστά ανώτερα αυτά του χρέους. Μόνο έτσι. Ε, και φυσικά να υιοθετήσουν δράσεις που θα, ενισχύει, θα ενισχύουν την ανάπτυξή τους. Ο κύριος Μαρτουσέλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Bloomberg πριν από κάποιες ημέρες ε, ε, δημοσίευσε μια μυστική επιστολή της Bank of Italia στο Αποπτικό Συμβουλίο της ΕΚΤ και εκεί γίνεται λόγος για τον κίνδυνο που υπάρχει να λαμβάνονται αυθαίρετα και αδικαιολόγητες αποφάσεις ε, διότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα των περιουσιακών στοιχείων και αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει αυτή η επιστολή και θέλω να μας αξιολογήσετε το γεγονός ότι πράγματι αυτό το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Και άλλη μία ερώτηση. Η Unicredit και η EMI στην Ιταλία, όπως γνωρίζετε, γνωστές εταιρείες ε, βρίσκονται σε δυσκολία. Είναι και οι δύο πολύ γνωστές στην περιοχή του Βένετο. Έχουν πρόβλημα ανακεφαλαίωσης. Υπάρχει κάποιο μέλλον άραγε για τις μικρές, τις λαϊκές τράπεζες. Ο κύριος Ντράγκη, κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις διαρροές του Bloomberg ανεξάρτητα από που προέρχονται. Επιτρέψτε μου όμως να αναφέρω κάποιες σκέψεις μου σχετικά με την αντίδραση του Εποπτικού ε, Συμβουλίου σχετικά με το TREPS. Πρώτον, υπάρχει μια γενική συζήτηση και η συζήτηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν είναι ολοκληρωμένη και εντωμεταξύ θα ακουστεί η άποψη, μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η άποψη όλων των ενδιαφερομένων. Θα γίνουν προσαρμογές αν κριτεί απαραίτητο. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι παρεπιπτόντως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ε, για να ε, είναι η αντίδραση του Εποπτικού Συμβουλίου περίπου όπως και αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να δημιουργήσουμε μειονέκτημα ε, στις τράπεζες σε σχέση με άλλες τράπεζες που διέπονται από διαφορετικό δίκαιο. Τώρα, το ε, κεφάλαιο, το μέσο κεφάλαιο που απαιτείται είναι αν θέλουμε να υπάρχει ένα buffer zone πάει στο 55. Υπάρχουν τράπεζες για τις οποίες ε, αυτή η απέτηση για αύξηση του ελάχιστου κεφαλαίου μπορεί να είναι ένα κίνητρο για να καλύψουν αυτή την απέτηση. Βεβαίως οι τράπεζες διαφέρουν διότι είναι και διαφορετικό το σημείο κίνησης και το Εθνικό Εποπτικό Συμβούλιο ε, ίσως να μην είναι τόσο σκληρό όσο πρέπει να είναι τώρα. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, ε, διότι οι λόγοι γιατί ε, λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τρεις. Πρώτον, αξιολόγηση κινδύνων. Δεύτερον, ε, εναρμόνιση και τήρηση της Συμφωνίας Βασιλεία 3. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και άλλες ε, ε, προϋποθέσεις όπως το τίλακ, ε, ο λόγος μόχλευσης που έχουν συμφωνηθεί ε, στο σχετικό πλαίσιο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Κατά τα άλλα, οι περισσότερες τράπεζες έχουν επίπεδο κεφαλαίου που είναι πολύ πιο πάνω από αυτό που απαιτείται από τον μηχανισμό SSM. Άρα δηλαδή η απειλή ότι δίθεν αυτό θα μπορούσε να απειλήσει την ανάπτυξη δεν ισχύει ε, διότι σας είπα αυτές οι τράπεζες έχουν τεράστια κεφαλαιοποίηση. Με λίγα λόγια, επαναλαμβάνω αυτό που είχα και πριν. Το να υπάρχουν ισχυρέ τράπεζε, αυτό είναι πολύ καλύτερο για την ανάκαμψη από ότι αδύναμε τράπεζε. Κατόπιν τούτου η αντίδραση του Εποπτικού Συμβουλίου του να υπάρχουν ισχυρές τράπεζες, αυτό είναι πολύ καλό, ακόμα και αν οι τράπεζες ε, μεσοπρόθεσμα δεν έχουν αρκετά κεφάλαια και ενδέχεται πράγματι να υποστούν κάποιες αρνητικές συνέπειες. Πάντως, αν θέλετε αυτές τις ερωτήσεις μπορείτε να τις υποβάλλετε ε, με πολλές περισσότερες λεπτομέρειες στην επικεφαλής του μηχανισμού SSM όταν θα έρθει εδώ. Το θέμα είναι ότι αν μια τράπεζα λειτουργεί σωστά, αν έχει σωστή ανακεφαλοποίηση, ε, εάν η τράπεζα κατορθώνει να ανταποκρίνεται στους κινδύνους που την απειλούν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το μέγεθος από μόνο του δεν είναι ε, αναχαιτιστικός παράγων για τις τραπεζικές δραστηριότητες. Υπάρχουν ε, άλλα μεγέθη που παίζουν ρόλο. Οι συνθήκες και οι προποθέσεις δεν είναι πάντα ίδιες. Ο κύριος Φερνάνδες. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε κύριε Δράγκη που ήρθατε. Σίγουρα πολλές ε, ερωτήσεις προκύπτουν από την ε, ομιλία σας. Είπατε στην αρχή ότι οι αναταραχές, οι αναταράξεις του καλοκαιριού θα ε, απαιτήσουν περισσότερο χρόνο για να επανέλθουμε σε ένα πληθωρισμό γύρω στο 2% αν χρειάζεται περισσότερος χρόνος και δεν αναλυθούν μέτρα, τότε φαντάζομαι ότι το διάστημα που περίμενε η ΕΚΤ για να φτάσει ο πληθωρισμός στο 2% θα είναι μεγαλύτερο και παρόλα αυτά δεν σκοπεύετε να, να λάβετε κανένα μέτρο για να το επισπεύσετε. Γιατί. Δεύτερον, για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών και τη ροή χρηματοδότησης από τις τράπεζες ε, προς σκιώδης, ε, το σκιώδης τραπεζικό σύστημα ή προς μη, ε, προς μη τραπεζικά ιδρύματα. Βλέπω μια μετατόπιση της ροής χρηματοδότησης προς μη τραπεζικά ιδρύματα. Όπως είπατε όμως, αυτά οι μη τράπεζες, non-banks, εκπίπτουν του, της της εποπτείας της ΕΚΤ. Γιατί δεν είναι τράπεζες. Οι τράπεζες εμπίπτουν στην εποπτεία της ΕΚΤ. Φυσικά θέλουμε να προωθήσουμε την Ένωση Κεφαλαγορών, αλλά δημιουργείται κίνδυνος ε, γιατί όλο και μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότησης ε, προέρχεται από διάβλους που εκπίπτουν ε, τις άμεσες εποπτείες της ΕΚΤ. Επίσης, στην έκθεση των πέντε προέδρων, στο δεύτερο στάδιο, μιλούμε για ένα αντικυκλικό μηχανισμό. Ερωτώ λοιπόν, αυτός ο αντικυκλικός μηχανισμός θα μπορούσε να είναι μία ασφάλεια για την ανεργία. Ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, θεωρούμε ότι η ποσοτική μας χαλάρωση ήταν αποτελεσματική και είχαμε βελτίωση στην Ευρωζώνη, κυρίως στις αγορές των τραπεζών και στον τραπεζικό κλάδο. Και είχαμε και κάποιες βελτιώσεις ε, ε, λιγότερες και στην αγορά εργασίας. Βέβαια αυξήθηκε ο κίνδυνος μείωσης του πληθωρισμού και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς όλους αυτούς τους κινδύνους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι έτοιμο, πρόθυμο και ικανό να αναλάβει δράση αν παραστεί ανάγκη. Και είπα ότι μπορεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσής μας να παραταθεί και μετά το Σεπτέμβριο ή να τύχει κάποιες προσαρμογής ως προς το μέγεθός του, τη σύνδεσή του και το σχεδιασμό του. Και μάλιστα απόδειξη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι έτοιμο να προσαρμόσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ανάλογα με τις εξελίξεις. Απόδειξη λοιπόν της ετοιμότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να αναθεωρήσει το πρόγραμμα ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του ήταν η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο ε, να περάσει το όριο έκδοσης από το 25% στο 33%. Επίσης, ε, η Ένωση Κεφάλαιο Αγορών και να είμαι σαφής καταρχήν. Το γεγονός ότι κάποιες ε, δραστηριότητες διαμεσαλάβησης ε, μετατοπίζονται από το τραπεζικό σύστημα σε μη τραπεζικά ιδρύματα δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική εξέλιξη. Είναι εν και φυσιολογική, γιατί έχουν απομοχλευτεί οι τράπεζες σε μεγάλο βαθμό, οπότε άλλα, άλλα ιδρύματα και αναλαμβάνουν αυτό το τμήμα που άφησαν οι τράπεζες. Και αυτό είναι θετικό, γιατί δεν θα στηριζόμαστε μόνο στις τράπεζες. Θα στηριζόμαστε όλο και περισσότερο στις αγορές γιατί η αποκλειστική εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό τελικά εμπόδισε την ταχύτερη ανάκαμψή μας το 2011 και το 2012. Οπότε αυτή η μετατόπιση είναι θετικό στοιχείο. Βέβαια, όσο αυξάνει ο σκιώδης τραπεζικός κλάδος, οι μη τράπεζες, υπάρχουν και κίνδυνοι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ή να αντιμετωπιστούν και με μακροπροληπτικούς μηχανισμούς. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε εποπτικό μηχανισμό και για μη τράπεζες ή για σκιώδες τραπεζικό σύστημα και κυρίως ε, για ε, ιδρύματα της αγοράς ή φορείς της αγοράς. Ευχαριστώ. Κύριος Ρωσάτη. Ευχαριστούμε κύριε Ντραγκή που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τη λειτουργία του ίστα του ε, δανειστή ε, ως λειτουργία της ΕΚΤ. Πέρυσι είχατε ανακοινώσει το πρόγραμμα για τις νομισματικές συναλλαγές και καταφέρατε να καθισχάσετε την κατάσταση στις αγορές χωρίς να ξοδέψετε ένα ευρώ. Ξέρω ότι αυτή η απόφαση δεν ληφθεί ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορείτε να αναλύσετε λίγο την επιχειρηματολογία ε, για ποιο λόγο η έκτησε μια νομισματική ένωση σαν τη δική μας ε, είναι καλό να λειτουργεί ο σύστατος ε, δανειστής ε, αφού, αφού τα επιχειρήματα κατά αυτού του ρόλου ακούγονται από τον πρόσωπο μίας μόνο τράπεζας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. I have a certain... Δυσκολεύομαι κάπως να απαντήσω αυτή την ερώτηση για μας και για μένα ο ίστατος ε, δανειστής αυτή η έννοια για τη, ε, για τη διακυβέρνηση για τις κυβερνήσεις ε, αυτό δεν επιτρέπεται από τις συνθήκες έχουμε το άρθρο 1.123 που απαγορεύει την παρακολουθή της χρηματοδότησης Γι' αυτό τα δύο προγράμματα OMT και QE επιτρέπουν όταν μια κυβέρνηση δεν έχει πρόσβαση στις αγορές ε, να αποτελεί το αντικείμενο μια ειδική εξαίρεσης και αγοράζουμε τότε τις ατομόλογα τη από τη δευτερεύουσα αγορά. Να διευκρινίσω την ερώτησή μου, λέει ο κ. Ροζάτη, δεν ήμουν σαφής. Αυτό που έλεγα ήταν η περίπτωση όπου έχουμε πανικό στην αγορά το οποίο ασκεί πίεση στα ομόλογα μιας χώρας που κατά βάση είναι φερέγγια αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες ρευστότητα. Μπορεί να έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου σε μια χρηματοπιστωτική αγορά να έχουμε ε, αυτή την, κακή ισορροπία. Τι ρόλο παίζει τώρα η ΕΚΤ εντός της Νομισματικής Ένωσης ώστε να αντιδρά προληπτικά να μην επιτρέπει να δημιουργηθεί τέτοιο ε, κακή ισορροπία. Αυτό που κάναμε σε εκείνη την περίπτωση τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, είναι έτοιμη να αγοράσει ομόλογα στη δευτερεύουσα αγορά της χώρας αυτής εφόσον η ίδια η χώρα ε, εφαρμόζει αξιόπιστες πολιτικές. Το λάθος είναι το να αγοράζει κανείς ομόλογα όταν οι πολιτικές ε, δεν είναι πιστικές, γιατί σε αυτή την περίπτωση αγοράζει έκτο όλα τα ομόλογα στην αγορά, διότι όλοι πολλούν τα ομόλογα, διότι ε, κανείς δεν εμπιστεύεται τις πολιτικές της χώρας. Ε, και γι' αυτό το λόγο εκείνη την εποχή η ΟΜΤ απέτησε η χώρα να ε, εγκρίνει συγκεκριμένα ε, προγράμματα χρηματοοικονομικής βοήθειας από το ESF και το IMF. Ε, είναι λοιπόν ίστατος δανειστής εντός των ορίων της αξιοπιστίας των οικονομικών πολιτικών της χώρας και στα πλαίσια πάντα της συνθήκης. Thank you, Kostas Ευχαριστώ, Κώστας Μαυρίδης. Incidentally, incidentally, uh, the συγγνώμη να πω και κάτι άλλο περιπτώντος ναι, δεν χρειάζεται βέβαια να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι η συμμόρφωση των πολιτικών ΟΕΜΤ με τη συνθήκη έχει ε, επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τράγκε, όσον αφορά στην ε, ερώτηση σχετικά με το μηχανισμό ΕΛΑ για την περίοδο 12-13, κυρίως ε, σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, νομίζω η σωστή ερώτηση είναι η εξή. Τελικά, ποιος είχε την νομική ευθύνη για την απόφαση που ελήφθη τότε. Ήταν η Εθνική Εποπτική Μονάδα ή η απόφαση ελήφθη από την ΕΚΤ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ελήφθη, ας πούμε, από τη Λαϊκή Τράπεζα τότε ή από την ΕΚΤ. Τώρα, στις 14 Σεπτεμβρίου, πριν από δύο μόνο εβδομάδες, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, ο κύριος Κωνστάντσιο, απάντησε σε μία ερώτηση του Reuters σχετικά με, τις, με την ελληνική κρίση με τον εξή τρόπο και παραθέτω, διαβάζω. Από πλευράς νομικής καμία χώρα δεν μπορεί να εκδιωχθεί ποτέ δεν τέτοιο ενδεχόμενο. Ισχύει λοιπόν αυτό ή όχι. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Σε τελική ανάλυση, ε, αυτά με την Ελλάδα ήταν μια έντιμη συμφωνία ή ήταν μια μπλόφα. Και, επειδή έχω και χρόνο, σχετικά με την έκθεση των πέντε προέδρων. Μερικοί εξημών, κύριε Ντράγκη, μερικοί λοιπόν εξημών είναι πεπισμένοι για τις ε, ισότιμες ευκαιρίες ε, και πιστεύουν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μας προσφέρουν την απαραίτητη προστασία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι με αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων αυτό θα έπρεπε να έχει εκπονηθεί εδώ και πολύ καιρό και ελπίζουμε αυτή τη φορά να μάθαμε από την κρίση Θέλω να το πιστεύω αυτό για την ΕΚΤΕ. Έχω και ένα παράπονο που θέλω να εκφράσω. Ξέρετε την προηγούμενη φορά όταν είχα την ευκαιρία να μιλήσω σας έκανα μια ερώτηση μέσω του Προέδρου και ξέρετε κάτι μου στείλατε απάντηση για λάθος ερώτηση. Τώρα αν θέλετε ε, δώστε μου ε, μια σωστή απάντηση για να μην είμαι πάλι την επόμενη φορά εδώ και να σας ξανακάνω τις ίδιες ερωτήσεις. Ο κύριος Τράγκη, λυπάμαι πολύ αν έγινε αυτό. Πάντως να σας πω κάτι, δεν ήταν σκόπιμο αν έγινε. Τώρα, η απάντηση είναι η εξής. Τότε στην Κύπρο η αρμόδια εποπτική αρχή η οποία θα έκανε την αξιολόγηση φερεγγιότητας ήταν η Εθνική Τράπεζα της Κύπρου. Σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είχαμε τη σύσταση εντωμεταξύ του SSM, του Μηχανισμού Διάσωσης, και ο μηχανισμός αυτός έγινε ε, εποπτική αρχή, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός έγινε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως και οι εθνικές τράπεζες είναι πολύ σημαντικές και εξακολουθούν να δίδουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη ρευστότητα των τραπεζών. Όμως η πραγματική αξιολόγηση στην οποία βασίστηκαμε εμείς, δηλαδή το Συμβούλιο της ΕΚΤ, αυτή η απόφαση ήρθε από το μηχανισμό SSM. Αυτά για την πρώτη σας ερώτηση. Τώρα, για την δεύτερη σχετικά με αυτά που είπε το μέλος του ε, Διοικητικού Συμβουλίου σε απάντηση στο Reuters, εγώ θέλω απλά να επαναλάβω η ΕΚΤ δεν είναι ο θεσμός εκείνος που αποφασίζει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Η ΕΚΤ ανέκαθεν λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί πάνω στην παραδοχή ότι όλα τα κράτη-μέλη θα παραμείνουν μέλη. Τώρα, ε, κατά πόσον αυτό είναι νόμιμο ή όχι, δεν θα τοποθετηθώ επ' αυτού, γιατί δεν ξέρω κιόλα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε στο τέλος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, και είναι και σημαντικό να γνωρίζουμε, ε, όπως και εσείς είπατε, να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους. Παρεπιπτόντως, όπως σας είπα και προηγουμένως, συστήσαμε τον οργανισμό, το μηχανισμό με συγχωρείτε SSM και τον SRM, όπως και το ε, Διοικητικό Συμβούλιο του SRM, άρα δηλαδή όλες τις τράπεζες και τους τραπεζίτες τους αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί να μην πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο και καταθέτες. Έχω λίγα δευτερόλεπτα στην ερώτησή μου κύριε Ντράγκη. Τα έχω μπερδέψει παρόλα αυτά. Τελικά για τον μηχανισμό έλα ποιο είχε την ευθύνη, η ε, τοπική εθνική τράπεζα ή η ΕΚΤ. Η απόφαση για τον ΕΛΑ είναι μια απόφαση που λαμβάνεται από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, η αξιολόγηση φεργιότητας στην περίπτωση της Κύπρου έγινε από την Εθνική Τράπεζα της Κύπρου στην Ελλάδα όμως. Σας είπα να ξύχαμε τον SSM και η αξιολόγηση έγινε από τον SSM. Όμως η απόφαση για τον ΕΛΑ εξακολουθεί να είναι προνομία της Εθνικής Τράπεζας μιας χώρας. Βεβαίως η ΕΚΤ μπορεί να μην ανταποκριθεί στο αίτημα. Δύο ερωτήσει. Ε, μπορούμε ακόμη να δεχτούμε. Αλλά επειδή πριν μπέρδεψα τον υπολογισμό του χρόνου, θα δώσω το λόγο σε, στον κύριο Ουρτασούν για μια δευτερολογία. Ε, ο ενίο υποπτικό μηχανισμό είπε για την Ελλάδα ότι ήταν αφαιρέγγυε σε τράπεζες. Ενώ είπατε ότι έγινε μια πιο δυναμική αξιολόγηση από την Κεντρική Τράπεζα για τι ασφάλειε. Αυτό δεν συνέβη στην Κύπρο, το κάνατε μόνο για την Ελλάδα. Γιατί λοιπόν αναπόκειται στη διακριτική σα ευχαίρεια τελικά. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Η απόφαση για τον ΕΛΑ επαφείται στη διακριτική σας ευχαίρεια, αυτό φαίνεται από τις δράσεις σας. Όχι καθόλου. Στην Κύπρο, η, η Κύπρος τηρούσε το σύστημα προσαρμογής, είχε δεχτεί το μνημόνιο, εφαρμοζόταν η πολιτική. Μπορούμε να το ελέγξουμε αν θέλετε. Η δυναμική αξιολόγηση που κάνουμε στηρίζεται στο γεγονός ότι βλέπουμε τις μελλοντικές εξελίξεις υπό το πρίσμα της βελτίωσης της αξίας των ασφαλιών, κάτι που δεν ίσχυε για την Ελλάδα. Ενώ ίσχυε στο παρελθόν. Οπότε αν το λάβετε αυτό υπόψη, διαπιστώνετε ότι οι αποφάσεις για τον ΕΛΑ είτε γινόταν από την, αρμό... για την εξολόγηση αρμόδιας εποπτικής αρχής και ή όταν δινόταν και δυναμική αξιολόγηση από την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις οδηγούσαν σε αύξηση της αξίας των ασφαλιών, των εγγύσεων και άρα ήταν υπέρ της φερεγγιότητας της τράπεζας. Επιχείρημα υπέρ της φερεγγιότητας. Τέλος, δεν έχετε δικαίωμα για συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Ουρτασούν. Να απαντήσω, μα θέλετε. Αν μια δυναμική αξιολόγηση δεν χρειάζεται, ε, και χρειάζεται μόνο μία αξιολόγηση χρόνου και χώρου. Εντάξει, αλλά όταν χρειάζεται μια δυναμική αξιολόγηση αφορά τι μελλοντικέ εξελίξει. Το κατά πόσο οι εξελίξεις βελτιώνουν την αξία των ασφαλιών, των εγγύσεων ή ε, την μειώνουν. Γιατί αυτό καθορίζει τη συνολική αξιολόγηση της Δεν είναι πολιτική εκτίμηση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το λόγο. Δύο ερωτήσει. Όσον αφορά από όσο μαθάμε στο Κοινοβούλιο, οι Εθνικές Αρχές της Ιταλίας σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας τράπεζας υπό το δικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν πράξεις εξυγένσης. Εσείς ε, συμμερίζεστε αυτή την ε, επιλογή της Υπουργού δεδομένου ότι και μέσω του SRM είναι δυνατόν να δοθούν τέτοια δεδομένα. Είναι σωστή αυτή η μέθοδος. Τώρα για το roadmap των πέντε προέδρων έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο B, διότι από ό,τι είπα ε, χθε σε μια κρόση ο Σόιμπλε, μιλώντας για το υποθετικό σενάριο μιας ε, ε, αναγκαίας ε, δημοσιονομικής ένωσης ώστε να λειτουργεί σωστά η νομισματική ένωση. Ε, αυτό το δημόσιο country by country reporting είπε ο ίδιος ότι το δικό του κοινοβούλιο ήταν αντίθετο. Ενώπιον λοιπόν αυτών των εθνικών αρχών μιας χώρας όπως η Γερμανία τέτοιες δηλώσεις Αξίζει να συνεχίσουμε να πιστέψει ο κόσμος αυτή την έκθεση των πέντε πρόεδρων ή όχι. Διότι διαφορετικά πρέπει να βρούμε ένα εναλλακτικό σχέδιο με ένα πιθανό ε, σενάριο εξόδου από το ευρώ μιας χώρας διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ε, ώστε να διατηρήσουμε και την νομισματική κυριαρχία των χώρο μας. Ευχαριστώ, αλλά ξέρετε δεν είναι εταιρεία με μετοχές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ένωση χωρών και πολιτών. Λοιπόν, για την πρώτη σας ε, ερώτηση δεν έχω απάντηση γιατί δεν γνωρίζω τίποτα. Για τη δεύτερη ερώτηση, όχι δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Αυτός είναι ο δικός χάρτης. Και βασίστηκε σε συζητήσεις και αποφάσεις και διαβουλεύσεις των ε, κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα κράτη-μέλη θα χαράξει το δρόμο όσον αφορά τις λεπτομέρειες του. Ευχαριστούμε και Σουέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ Πρόεδρε Εντράκη που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Σημείωσα κάποια από τα σχόλια που ακούσαμε νωρίτερα και βασίστηκαν ε, στην εκθέση των πέντε Πρόεδρων και τις παρατηρήσεις σας σήμερα για την ανάγκη πιο ολοκληρωμένης ένωσης ε, για την Ευρωζώνη και πολιτικές ε, κατάλληλες δράσεις ε, για ολόκληρη την Ευρωζώνη ώστε αυτή να γίνει πιο νευμερή καλύτερα. Μπορείτε να μου πείτε κάποιες ιδέες πώς θα εξασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη στη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης μαζί με την δικαιοσύνη στη διακυβέρνηση ε, στην ε, ενιαία αγορά που, για τα μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Είναι σημαντικό ζήτημα και πρέπει να μην το ξεχνάμε. Αφενός τα μέλη της Ευρωζώνης θέλουν να έχουν την ελευθερία να εντείνουν την ολοκλήρωση, να την προχωρήσουν όπως απαιτείται όταν κάποιος έχει κοινό νόμισμα. Η ύπαρξη κοινού νομίσματος συνεπάγεται κοινέ ευθύνε, ε, λήψη κοινών αποφάσεων σε πολλούς τομείς. Είναι μια διαδικασία πιο εκτενής ε, από αυτή που αφορά τα χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ μη μελών και μελών, ώστε τα μέλη να μπορούν να είναι ελεύθερα να συνεχίσουν να προχωρούν προς μια πιο τέλεια ένωση. Ταυτόχρονα τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν συναισθηθεί το γεγονός ότι υπάρχουν συμφέροντα που αφορούν αποκλειστικά τα μη μέλη και πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη. Το πιο σημαντικό από τα οικοδοματά μας που πρέπει να ε, διατηρηθεί και να βελτιωθεί είναι η νέα αγορά. Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις από τα μέλη της Νομισματικής Ένωσης μπορούν να είναι επικοδομητικές, θετικές, ε, να υποστηρίξουν την ενιαία αγορά και την πρόοδο της ενιαίας αγοράς. Ξέρουμε ακόμα ότι χρειάζονται πολλά βήματα να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο Ντράγκη, όλους σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική η ανταλλαγή απόψεων εδώ. Ο επόμενος νομισματικός διάλογος θα λάβει χώρα 12 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, Παρακαλώ, καθίστε κύριε και κύριοι. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. is... Επόμενο σημείο τη διάταξη είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπή ΕΚΟΝ επί τη εκθέσεως που έχει τίτλο Οδεύοντα προ μία ενιαία ψηφιακή αγορά αρμόδια για την εκπόνηση της Επιτροπής αυτής είναι η Επιτροπή ΙΜΚΟ. Εμείς απλώς γνωμοδότηση θα συντάξουμε. Ο κύριος Ρένατος Σόρου είναι ο εισηγητής μας, ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Θα πρότεινα λοιπόν να, να περάσουμε στη συζήτηση. Θα δώσω τέσσερα λεπτά στο συντάκτη της γνωμοδότησης και τρία λεπτά στον κάθε σκιώδη. Έχετε το λόγο κύριε Σόρο. Εδώ και καιρό συζητάμε για το πώς θα δώσουμε μεγαλύτερη έθωση στο ψηφιακό τομέα στην Ευρώπη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες όλο και περισσότερο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, του τρόπου ζωής, του τρόπου διαχείρισης των πραγμάτων. Είναι κυρίαρχο κομμάτι στην κοινωνία μας. Πολλά έχουν να γίνουν και πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθούν οι υποδομές δικτύων και πολλές ε, περιοχές της ε, Ευρώπης ε, ε, δεν έχουν επαρκή δίκτυα, επαρκείς υποδομές ε, για να μπορέσουν να στηρίξουν αυτό το σημαντικό τομέα. Οι ικανότητες επίσης, ε, οι τεχνικές ικανότητες και γνώσεις στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας δεν είναι επαρκή ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία 100%. Και επίσης πρέπει να υπενθυμίσουμε σε αυτή την Επιτροπή ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κυριαρχούν στην αγορά των τεχνών, των καλών τεχνών ε, και των ψηφιακών ε, πλατφορμών ε, βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γι' αυτό χαίρομαι για το σχέδιο δράσης της Κομισιόν για την ψηφιακή ενιαία αγορά που δημοσιεύτηκαν σχέδιο το οποίο προσπαθεί να δώσει μια απάντηση σε αυτές τις καθυστερήσεις, σε αυτές τις ευθύνες, σε αυτές τις δράσεις που απομένουν να ολοκληρωθούν. Απομένει να δούμε ποιες ε, ε, δράσεις πραγματικά θα υλοποιηθούν. Η έκθεση για αυτό το σχέδιο δράσης ε, αναθέτει στην Ήτρε και στην Ίμκο και στη δική μας Επιτροπή την ιδιαίτερη ευθύνη της ε, διασυνοριακής φορολογίας. Πολύ σημαντική όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικό εμπόριο που υπολογίστηκε ότι οι επιχειρήσεις μας οι οποίες έχουν να κάνουν με 28 διαφορετικότητα ΦΠΑ στην Ευρώπη ε, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας ε, και δεν μπορεί η αγωνιστικότητά τους να υπονομεύεται όταν έχουν να κάνουν με άλλες χώρες. Είναι σημαντικά ζητήματα που άρχισαν να συζητώνται χθε στην ε, Επιτροπή Τάξη, όπου συμμετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών. Στις 1.500 ε, ε, προτάσεις που προβλέπονται στην έκθεση, εστιάζομαι σε τρία σημεία. Στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές στην Ευρώπη σε επαρκές επίπεδο. με αυτό ασχολήθηκε και το σχέδιο Juncker. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση πριν από ένα χρόνο και ακόμα σήμερα δεν έχει φτάσει τίποτα από τελικές αποφάσεις και σε επιχειρήσεις το οποίο θα μεταφραζόταν σε επενδύσεις. Επίσης το ψηφιακό χάσμα δεν θα έπρεπε να διαφοροποιεί τις περιοχές μας, θα έπρεπε να οδηγεί σε επενδύσεις ε, στην ψηφιακή τεχνολογία ώστε να επιτευχθεί ε, αυτή η διαδικασία σύγκλησης. Και τέλος προσπάθησα να υπογραμμίσω τις ε, πτυχές της πολιτικής ανταγωνισμού. Τομές που έχει ιδιαιτερότητες. Τα δίκτυα τείνουν να αναπτύσσονται και να εμποδίζουν την γέννηση άλλων δικτύων. Κάθε επιπλέον ε, στοιχείο δικτύου προσθέτει αξία στα προηγούμενα δίκτυα. Σε αυτό προστίθεται ότι στην ψηφιακή οικονομία υπάρχει και το οριακό κόστος μηδέν. Το ουσιαστικά είναι πολύ ανταγωνιστικές ε, οι οικονομίες αυτές ε, σε σχέση με τις επιχειρήσεις μας. Έχουμε νέα πλατφόρμες που αρχίζουν να μονοπολούν την οικονομία. Και όλοι θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας αυτό και να βρούμε διορθωτικά μέτρα. Αυτά τα σημεία προσπαθώ να υπογραμμίσω στις 1500 προτάσεις μου. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους σκιώδεις ηγητές. Εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Πέλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.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 Η οικονομία αυτή ε, έχει τεράστιο δυναμικό και μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχω τρία λεπτά στη διάθεσή μου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει συντονισμός μέσω του προγράμματος στρατηγικών επενδύσεων και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι ο τομέας αυτός ε, συνεχίζει να αναπτύσσεται και χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που να οδηγεί στην ανάπτυξη. Εγώ συμφωνώ με αυτό το έγγραφο και πράγματι είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται οι διάφοροι φορείς, ε, κυρίως ε, Όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουμε περαιτέρω αναπτυξιακό δυναμικό. Λοιπόν, ακράταντα πεπισμένος ότι ε, μια καλά οργανωμένη ψηφιακή αγορά ε, μπορεί να συμβάλλει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και υπάρχουν δυστυχώς και πολλά κενά θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα προβληματικό τομέα, διότι το σημείο 4 σαφώς ε, και είναι σημαντικό, ε, πρόκειται για φορολόγηση και είμαι πεπισμένος ότι μια ψηφιακή εσωτερική αγορά ε, χωρίς τη σωστή φορολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Υπάρχουν ε, ε, ανομαλίες ε, στα λογιστικά, αλλά θεωρώ ότι αυτά όλα είναι και θέμα κυβερνήσεων. Εδώ πρόκειται ξεκάθαρα για δημοσιονομικές επιπτώσεις, άρα δηλαδή χρειαζόμαστε συμβιβασμούς. Σε γενικές γραμμές, εν πάση περιπτώσει, μπορώ να σας πω ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι ένα πολύ καλό σημείο κίνησης και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως και θα είχα να κάνω και άλλες συμπληρωματικές προτάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοδομητική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των μεταρρυθμιστών συντηρητικών για τρία λεπτά, κυρία Σουίνβερ. Ευχαριστώ. Η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι ένα τομέα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής, κυρίω για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν χρειάζονται πια δαπανηρέ υποδομές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά ε, και φτάνουν σε πελάτες και πέραν των χωρών του. Το θέμα είναι με τον κανονισμό ε, το κανονισμό μας είναι ε, και δεν ανταποκρίνεται στο τεράστιο δυναμικό τη ψηφιακή αγορά. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα προσαρμόσουμε τους κανόνες για να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και να μην δημιουργήσουμε νέους ε, περιττούς διασυνοριακούς φραγμούς στην ψηφιακή εποχή. Ο κύριος Σόρου αναφέρεται στην εναρμόνιση του κανονισμού για το crowdfunding. Ε, είναι σημαντικό, αλλά να δούμε το θέμα της προστασίας των καταναλωτών, γιατί κάποιες πλατφόρμες ε, για τέτοιο έρανο crowdfunding ε, θυμίζουν ε, ε, κάποιες πλατφόρμες επενδυτικές και δεν καλύπτονται από την προστασία της οδηγίας MIFID. Βέβαια είναι σημαντική πηγή εισόδων, εσόδων μάλλον για επιχειρήσεις που αλλιώς θα πάσχιζαν, αλλά θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τους πιθανούς επενδυτές για τους κινδύνους, γιατί μπορεί έτσι να χάσουν όλες τους τις επενδύσεις. Ίσως προς το παρόν αυτό είναι αρκετό. Δεν πιστεύω ότι η εναρμόνιση διεξοδικών διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή σε μια πλατφόρμα που βρίσκεται μόλις στα Σπάργανα. Ίσως καλύτερα να επικεντρωθούμε στην προστασία του καταναλωτή προς το παρόν και πέραν του crowdfunding. Ε, θα θέλαμε στη γνωμοδότηση μας να δούμε τις νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, fintech που υπάρχουν. Η τεχνολογίες ε, οι νέες χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν ε, εικονικά νομίσματα όπως το bitcoin και χρησιμοποιούνται όχι μόνο για πληρωμές αλλά και για μεταεμπορικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα διακανονισμό τίτλων και χρεογράφων και ίσως ε, δημιουργήσουν επανάσταση στην όλη ψηφιακή αγορά και μειώσουν το κόστος των επενδυτών. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε αυτές τις νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, τις FinTech, αλλά ταυτόχρονα η, να μην τις εμποδίσουμε με τους ε, υφιστάμενους κανονισμούς. Θα πρέπει να δούμε το CSDR και την οδηγία MIFID, ώστε να δώσουμε ευκαιρία και σε αυτές τις καινοτόμες ε, χρηματοοικονομικές τεχνολογίες να δραστηριοποιηθούν και να ανθίσουν. Ε, για παράδειγμα, είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, μία καινοτόμη δραστηριότητα και τη Sunbox Approach. Να δούμε πώς οι φυστάμενοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν στις νέες επιχειρήσεις και πώς θα πρέπει αυτές να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή της ψηφιακής αγοράς που διανύουμε. Θα μπορούσατε μήπως στη γνωμοδότησή σας να συμπεριλάβετε και αυτές τις νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, τις FinTech. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόρβαλτς από τους φιλελεύθερους κανονικά είναι στο κατάλογο, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Μήπως τον αντικαθιστά κάποιος άλλος από τους φιλελεύθερους. Όχι. Οπότε ο κύριος Μίσο Ρέιμαν από τους πράσινους ή κάποιος άλλος τέλο πάντων από τους πράσινους αλλά δεν βλέπω κανέναν σκιώδη από τους πράσινους και οι FTD έχουν εκπρόσωπο ποιος θέλει το λόγο για τη γνωμοδότηση του κύριου Σόρου. Η ΕΝΕΦ, καδινήσει το λόγο από το κόμμα ΕΝΕΦ. Όχι, οπότε περνάμε στους λοιπούς ευρωβουλευτές. Θέλει κανείς το λόγο. Η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που έχασα την αρχή της συζήτησης και ζητώ συγγνώμη κύριε Σόρου. Σύμφωνο με τα όσα είπαν οι υπόλοιποι, είναι σημαντική η τομή σε αυτή. Ε, μια επιφύλαξη που έχω εγώ για την οποία θα υποβάλω τροπολογίες είναι το ζήτημα της εισαγωγής νέων φορολογικών συστημάτων που εισήξαν στην ψηφιακή η αγορά και πιο συγκεκριμένα το νέο σύστημα ΦΠΑ το οποίο ενώ βασίζεται σε σωστά κίνητρα για να αποφεύγεται η φορά αποφυγή πολυεθνικών που ε, αλλάζουν ε, θέσεις στις ε, δραστηριότητες τους για καλύτερα ποσοστά ΦΠΑ. Το νέο σύστημα δεν βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το αντίθετο, για πολλές στη δική μου χώρα, πολλές χρειάζεται να κλείσουν. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Συγητή συγγνώμη και αν θα είχε την ε, καλοσύνη να δεχθεί κάποιες ε, τροπολογίες. Ειδικότερα ο Επίτροπος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο Επίτροπος Άνσιπ, είπε ότι θα δημιουργήσει ένα κατόφλιο για τις εταιρείε αυτές ε, στο πλαίσιο του καθεστώτος ΦΠΑ, αλλά δεν μας είπε πότε. Αυτές οι ψηφιακές εταιρείε κλείνουν λόγω αυτού του προβλήματος και ελπίζω ο εισηγητής να μπορέσει να δεχθεί κάποιες τροπολογίες επί του ζητήματος. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να ζητήσω από τον κύριο Σίγητη, αν επιθυμεί να προσθέσει κάτι σε αυτή τη φάση της συζήτησης. Κύριε Σόρου, ναι, 30 δευτερόλεπτα για να καθισκάσω τους συναδέλφους. Ναι, θα φροντίσω να λάβω υπόψη όλα τους τα σχόλια και αν έχουν χρόνο θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια συζήτηση ώστε να τα εξετάσουμε όλα από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να σας ενημερώσω ότι οι επιτροπές ΙΜΚΟ και οι ΤΡΕΣ συνεργάζονται για την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης για τον κανόνα 55. Τελική ψηφοφορία για αυτή τη γνωμοδότηση σε αυτές τις επιτροπές θα λάβει η χώρα 20 Δεκεμβρίου. Όσον αφορά το δικό μας χρονοδιάγραμμα για αυτή τη ε, γνωμοδότηση, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 15η Οκτωβρίου, εξέταση των τροπολογιών 30 ε, Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 1η Δεκεμβρίου, ψηφοφορία ε, στις ε, λοιπές επιτροπές στις 10 Δεκεμβρίου και τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια κάποια στιγμή τον Ιανουάριο του 2016. Uh, Περνάμε στο, τελευταίο, στο πραγματικά τελευταίο σημείο της uh, ε, τη διάταξης, τα διάφορα. Υπάρχει κάτι που θέλουν να προτείνουν τα μέλη, δεν βλέπω τίποτα, οπότε δεν έχουμε κάτι επίγον, από ό,τι φαίνεται. Πριν κλείσω τη συνεδρίαση, να σας ενημερώσω για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα λάβει χώρα την 3η 13 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 και μετά συνεχίζουμε από τις 3 μέχρι τις 6.30. Αυτά για σήμερα. Κρίσω το τέλος της συνεδρίασης και σας εύχομαι καλό βράδυ.